Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίσατε θερμότατα ε, σε ένα αλλιόλουστο απόγευμα Δευτέρας. Παρ' όλα αυτά, η θέση μας εμάς εδώ είναι. Στην αίθουσα αυτή που τώρα ονομάζεται Αλτσίρτε Ντεγκάσπαρη, γιατί τη βαφτίσανε από την τελευταία φορά και όχι πλατεία Λουξεμβούργου δηλαδή γιατί δεν είμαστε στην πλατεία, αλλά είμαστε στη συνεδρίαση και χαιρόμαστε για την ημερήσια διάταξη που μας περιμένει. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνεται λοιπόν ούτως. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή για δύο δραστηριότητες που αποφασίσαμε εμείς οι ίδιοι. Η μία είναι στις 19 Απριλίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, η εκδήλωση με τα Εθνικά Κοινοβούλια με θέμα την κλιματική αλλαγή και την προστασία του κλίματος. Ελπίζω να είναι πολύ παρόντες και να συζητήσουν με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια για αυτό το μεγάλο θέμα και εν ώψη και της μεγάλης διάσκεψης για το κλίμα που επίκειται. Επίσης αποφασίσαμε να κάνουμε ένα εργαστήρι για την οδηγία σε Βέζο 3 αυτή την εβδομάδα, την Τετάρτη μεθαύριο στις 2 το απόγευμα με 6.30 στην αίθουσα Γιάν 6Q2 στον έκτο όροφο του παρόντος κτηρίου. Και θα χαιρόμουν πολύ να δω πολλούς συναδέλφους. Ζήτησε το λόγο Κριστέιβης, ορίστε παρακαλώ. Γενικά, θα ήθελα να πω ότι ε, ε να κάνετε ανακοινώσει του Πρόεδρου. Ξέρετε, οι πρόεδροι των επιτροπών ε, προέβησαν ε, σε ένα αίτημα στη διάσκεψη των προέδρων των πολιτικών ομάδων σε ό,τι αφορά ε, την νομοθεσία για διάφορους πίνακες που συμπεριλαμβάνονται στη νομοθεσία στην ε, οδηγία για την, ε, της Επιτροπής Γεωργίας υποστηρίξαμε μία πρόταση και σημειώσαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να ε, αντιπαρατεθούμε με το Συμβούλιο και ε, αντίστοιχα να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω ότι επίκειται έκθεση τώρα και ε, κάποιος εισηγητής ζητάει να διαγραφεί αυτό. Γιατί είναι πολιτικό αυτό το θέμα, θα μπορούσατε όμως να ζητήσετε από τη Γραμματεία να μοιράσει ένα σημείο μας στα μέλη της Επιτροπής και στους πολιτικούς συμβούλους να μας εξηγήσετε ποια είναι η σημερινή θέση της διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και των πολιτικών ομάδων για να μην καταντήσουμε τελικά στην Επιτροπή μας να ψηφίζουμε με τρόπο που αντιτίθεται στη συλλογική αντίληψη των ε, ηγετών μας και των Πρόεδρων των πολιτικών ομάδων. Καλώς. Αύριο το δουν οι συντονιστές αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Και θα έχουμε ευρύτερο φάσμα και πιο διαφανή συζήτηση. Καλωσορίζω θερμότατα ε, στην Ομιγύρη την κυρία Σοφία Κονή. Καλημέρα σας νέο μέλος, διότι η κυρία Σουή επέστρεψε ε, στη Γαλλία και τώρα είστε εσείς μέλος αυτής της ωραίας Επιτροπής Περιβάλλοντος. Καλώς και καλή επιτυχία στο έργο σας και καλή δύναμη. Έρχομαι λοιπόν στο σημείο 3 τώρα. Έγκριση των πρακτικών της 7 Μαρτίου και της 24ης, 25ης, 26ης Ιανουαρίου και όπως πάντα αν δεν έχετε επιφυλάξεις ε, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Ερχόμαστε στο σημείο 4 λοιπόν. Θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση αποβλήτων στους συντονιστές είχαμε πει ότι θα καλούσαμε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα μαζί της και θα δώσω το λόγο στην κυρία Σολεδάδ Μπλάνκο, Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, για να μας παρουσιάσει το θέμα. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Chairman, and thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ε, Επιτροπή σας για την πρόσκληση που απέστειλε στην ε, Επιτροπή να παρουσιάσει αυτές τις ε, τις θεματικές και τη στρατηγική και τη διαχείριση των αποβλήτων. Η έκθεση αυτή ε, υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και διαβιβάστηκε στα άλλα όργανα. Πρόκειται για μια στρατηγική η οποία υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2005 σαν μία από τις πέντε στρατηγικές που προήλθαν από το έκτο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης. Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος και στρατηγικής ήταν να προσανατολιστεί η Ευρώπη προς μια Ευρώπη της ανακύκλωσης και μιας πιο ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων και των απορριμμάτων. Η έκθεση που έχετε μπροστά σας είναι μια σύνοψη των κυριότερων δράσεων που ανέλαβε η Επιτροπή για να υλοποιήσει αυτή τη στρατηγική το δεύτερο, στο δεύτερο τμήμα γίνεται μία ανάλυση για τον αντίκτυπο της στρατηγικής αυτής, τόσο στην παραγωγή όσο και στη διαχείριση των αποβλήτων και τέλος υπάρχουν συστάσεις για μελλοντικές δράσεις. Υπάρχει φυσικά, υπάρχουν φυσικά και πολύ καλά στατιστικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων ε, στατιστικών στοιχείων ανά κράτος μέλος στο παράρτημα. Θα αναπτύξω εν συντομία το περιεχόμενο αυτών των τριών μερών που ανέφερα. Καταρχήν, σε σχέση με τις δράσεις που ήδη ανέλαβε η Επιτροπή για την υλοποίηση της θεματικής στρατηγικής για την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Από αυτήν την άποψη η Επιτροπή το 2005 από το 2005 και μετά έκανε πολλές προσπάθειες για την εναρμόνιση και την απλούστευση της νομοθεσίας που υιοθετήθηκε μετά από την ε, υιοθέτηση και την έγκριση της στρατηγικής. Το κύριο παράδειγμα είναι η υιοθέτηση το 2008 της αναθεωρημένης οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα, η οποία απλοποίησε και διευκρίνησε ε, τη γενικότερη πολιτική της Ένωσης. Ε, η οδηγία αυτή εγκαθιστά μια υποχρεωτική ιεραρχία και ε, ορίζει και την κατάρτιση στρατηγικών πρόληψης. Δημιουργήθηκε ένα κέντρο συλλογής στοιχείων για τα απόβλητα στην Eurostat και μία πλατφόρμα αναφοράς για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής αποφασίστηκαν ε, νέοι στόχοι για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα και συμπεριελήφθησαν στην αναθεώρηση της οδηγίας. Η πρώτη ανάγνωση έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται να ε, μπούμε στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης με σκοπό την έγκριση. Αν δούμε την πρόοδο που σημειώθηκε για την υλοποίηση της ιεραρχίας των αποβλήτων, Θέλω να κάνω μερικά σχόλια σε σχέση με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων. Για την παραγωγή απορριμμάτων και αποβλήτων. Η μείωση της παραγωγής ε, απορρίτων είναι ένας από τους στόχους της θεματικής στρατηγικής. Η έκθεση που εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούνιο δείχνει μια ανάμεικτη εικόνα. Σε γενικές γραμμές πρέπει να παραδεχθούμε ότι η παραγωγή απορριμμάτων αυξήθηκε σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά, και αυτό είναι το καλό, το θετικό, η αύξηση αυτή έγινε με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με την αύξηση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια συσχέτιση μεταξύ της συνολικής παραγωγής απορριμμάτων και της αύξησης του ΑΕΠ. Από το 2008 υπάρχει μια βραδύτερη μείωση, ωστόσο, την οποία πρέπει να την παρακολουθήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσο εκφράζει μια πραγματική τάση ή είναι απλώς αντανάκλαση της οικονομικής κρίσης, η οποία ξεκίνησε περίπου τότε. Η τάση η μείωση ή η αύξηση που είναι βραδύτερη από την αύξηση του ΑΕΠ αφορά όλες τις χώρες, ισχύει σε όλες τις χώρες. Αλλά όπως είπα τα αποτελέσματα διαφέρουν πάρα πολύ σε σχέση με την δημιουργία απορριμμάτων, για παράδειγμα μεταξύ των οικιακών απορριμμάτων. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των οικιακών απορριμμάτων αναέτος είναι λίγο λιγότερο από 500 κιλά, που αν το συγκρίνεις με τον αντίστοιχο μέσο όρο των Ηνωμένων Πολιτειών, 750, ε, είναι μεγάλη διαφορά, αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 300 κιλά μέχρι 800 κιλά. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για τη μείωση της ε, δημιουργίας αποβλήτων και απορριμμάτων. Μέχρι στιγμής όμως μόνο ένα κράτος, η Γερμανία, κατάφερε να μειώσει κατά 10% την παραγωγή οικιακών απορριμμάτων εντός της Γερμανίας. Όσο αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, γενικά η ανακύκλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε. Το 2008 η ανακύκλωση ήταν περίπου 13%, το οποίο δείχνει πρόοδο σε σχέση με το 2005, όταν ήταν μόνο 5, ήταν 5% λιγότερο και 18% όχι 80, 18% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό του 1995. Καλά νέα λοιπόν για την ανακύκλωση. Επίσης μειώθηκαν και μειώθηκε η χρήση του χώρου ταφής, υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Τώρα είναι 40% σε σχέση με 65% το 1995. Μειώσαμε λοιπόν από 65% στα 50% και στα 40% πιο πρόσφατα το ποσό των απορριμμάτων που πήγαιναν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Μερικά κράτη-μέλη έχουν εντελώς καταργήσει τις, τους χώρους υγειονομικής ταφής ε, στην επικράτειό τους, αλλά τα περισσότερα κράτη-μέλη βασίζονται στους χιτά, στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Αρχή, έχουμε ξεκινήσει να αναλύουμε ε, τις που οφείλονται οι διαφορές ε, αυτών των, σε αυτές τις επιδόσεις και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό οφείλεται σε ένα συνδυασμό μέτρων, κίνητρα, φορολογικά μέτρα, εκπαιδευτικά μέτρα, το σύνολο των πακέτων για μια κοινωνία της ανακύκλωσης. Όσο αφορά το μέλλον για τη διαχείριση των αποβλήτων, η έκθεση καταγράφει κάποιες τάσεις που πρέπει να μας καθοδηγήσουν στο μέλλον στην εκπόνηση της σχετικής πολιτικής. Πρώτον, ε, πρέπει να έχουμε αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, αποδοτική χρήση της ενέργειας και να χρησιμοποιούμε περισσότερα ανακυκλωμένα απόβλητα, έτσι ώστε τμήμα για, το τμήμα για την αυξημένη ζήτηση πόρων που είναι πολύ υψηλότερη αυτή τη στιγμή και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον σε σχέση με το παρελθόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι της ε, ανακύκλωσης αποβλήτων. Πρέπει να παράγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς και υλικά που βασίζονται σε ανακύκλωση προηγούμενων υλικών. Ε, πρέπει να υπάρχουν, υπάρχουν φιλόδοξοι στόχοι ε, για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό μπορεί να στηριχθεί να υποστηριχθεί από την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, η μείωση των χιτά, η αυξημένη ανακύκλωση και η μείωση της ε, εξάρτησής μας από την εγκατάλειψη απλώς των απορριμμάτων θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τις εκπομπές του δεξιού του άνδρακα για παράδειγμα. Τώρα, σε οικιακό επίπεδο, σε επίπεδο νοικοκυριού, ε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες εκεί για τη σημαντική μείωση των εκπομπών του, των αερίων του θερμοκηπίου με τη χρήση των περισσότερων ανακυκλωμένων υλικών. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των υλικών και των προϊόνων που επηρεάζουν όλα τα στάδια ζωής στο περιβάλλον. Και γι' αυτό ε, ενισχύουμε τις προσπάθειές μας, εντείνουμε τις προσπάθειές μας ε, για να αυξήσουμε τις γνώσεις μας και να μπορέσουμε να αριθμητικοποιήσουμε, να ποσοτικοποιήσουμε καλύτερα αυτόν τον αντίκτυπο. Όπως φαίνεται στην έκθεση, η υλοποίηση παραμένει υψηλή προτεραιότητα. Έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας να αυξήσουμε το επίπεδο υλοποίησης στα κράτη-μέλη, αλλά και πάλι το 2009 20% των συνολικών αγωγών ε, επί παραβάση του κοινοτικού δικαίου έχουν να κάνουν με τα απόβλητα και τα απορρίμματα. Δεν θέλουμε να βασιστούμε μόνο στην παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, στη διαδικασία επί παραβιάση του κοινοτικού δικαίου για να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να σημειώσουν πρόοδο, αλλά θέλουμε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις λύσεις που έχουν δώσει τα πιο προηγμένα κράτη-μέλη. Χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα λοιπόν, αλλά σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες έχουν να κάνουν και με τους λιγοστούς ε, ανθρώπινους πόρους που συμμετέχουν στον τομέα αυτό. Επιπλέον, εγκατακλείδη κύριε Πρόεδρε, οι κύριες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι να εδραιώσουμε ακόμα καλύτερα τις πολιτικές ανακύκλωσης και να, καταρ... και να αναπτύξουμε πιο στενές σχέσεις με τους άλλους τομείς πολιτικής. Προσπαθούμε να μεταφράσουμε αυτούς τους στόχους, αυτές τις προκλήσεις σε πρακτικές δράσεις, τις οποίες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά που θα πρέπει να αναλάβουν και τα κράτη-μέλη. Από τη μία πλευρά πρέπει να εντάξουμε καλύτερα την αποδοτική χρήση της ενέργειας στην πολιτική για τα απόβλητα και τα απορρίμματα και θέλω να πω ότι θα υπάρξουν πολλές πρωτοβουλίες ε, σε σχέση με τα απορρίμματα στο μέλλον σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης ε, θα υπάρξει όθηση και έμφαση στην πρόθεση και την πρόληψη. Υπάρχει ένα κεφάλαιο για την αποδοτική χρήση της ενέργειας στην έκθεση. Ε, εμείς στη Γενική Διεύθυνση ασχολούμαστε και με το θέμα των πρώτων υλών και επιδιώκουμε μια διεθνή συνεργασία πάνω στις πρώτες ύλες. Το 2014 θα έχουμε μια οδηγία πλαίση, την οδηγία πλαίσιο που θα αναθεωρηθεί και θα μας επιτρέψει ίσως να θέσουμε άλλους στόχους, πιο συνεπείς με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα παρακολουθήσουμε την υλοποίηση της οδηγίας πλαισίου και θα εκτελέσουμε και μια αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων διαχείρισης και πρόληψης θα εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι της Ένωσης ε, ότι οι πόροι θα δοθούν στα κράτη-μέλη και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές της ιεράρχησης των απορριμμάτων και των αποβλήτων. Αυτή ήταν μια πολύ μικρή σύνοψη του περιεχομένου της έκθεσης. Είμαστε στη διάθεσή μας να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μπλάνκο για την ε, παρουσίαση της έκθεσής σας. Όντως τα απόβλητα ε, είναι προτεραιότητα για μας ε, που ασχολούμαστε με την πολιτική περιβάλλοντος και βλέπουμε και πόσο συνδέεται αυτό με την κλιματική αλλαγή, την καταπολέμησή της και τα λοιπά. Τρεις έχουν στήσει το λόγο. Πρώτος ο Φλόρεντς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βγενέστατη ε, κυρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να διαφωνήσω σε δύο θέματα, να τη διαψεύσω. Ακούω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, υπάρχει πρόβλημα προσωπικού και για τον έλεγχο των ε, κανόνων που έχουμε ψηφίσει στην Ευρώπη δεν έχουν ούτε μια ντουζίνα υπαλλήλου. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να το διαχειριστεί από μόνη τη αυτό. Και δεύτερο, δέχομαι βεβαίω ότι το θέμα είναι δύσκολο και τα κράτη-μέλη ε, έχουν κάποια επιμονή ε, να αντιστέκονται στο να εφαρμόζουν μέτρα που τα ίδια τα κράτη έχουν ψηφίσει ε, στην Ευρώπη. Κατά τα άλλα, ομολογώ και εγώ και ότι παρακολουθώ την υπόθεση αυτή των θεμάτων του περιβάλλοντος εδώ και χρόνια και είναι πρώτη τάξεως αποτυχία αυτό που ζούμε σήμερα. Πρώτη τάξεως. Στα παλιά κράτη-μέλη οι διαφορές ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, ας πούμε, ή τη, Γαλλία και, τη Γερμανία και την Αγγλία είναι μεγαλύτερα μεγαλύτερες διαφορές από ό,τι μεταξύ Γερμανίας και Βουλγαρίας. Τα παλιά κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν την οδηγία πλαίσιο ε, ολιγορούν και όταν την εφαρμόζουν την οδηγία αυτή ε, χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες της παρόλο που ενημερώθηκε πριν από ε, δύο χρόνια οδηγία αυτή γιατί παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών ορισμός προτύπων και προδιαγραφών. Ξέρουμε στο Συμβούλιο ποιοι συνεδριάζουν χειροκρότησαν όλοι για τις πρώτες ύλε και είπαν ότι βεβαίως όλα αυτά είναι σημαντικά και θα πρέπει να προχωρήσουμε. Μετά από μία ώρα ο ίδιος υπουργός, μάλλον ε, ε, ε, το ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο ψήφισε για την οδηγία για τα 3 ε, τα ηλεκτρονικά απόβλητα και ο δικός μας υπουργό δεν έλαμψε εκεί με τη στάση του και πρόκειται για ευρωπαϊκούς κανόνες, απλούς κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουν λίγο τον εαυτό του στον τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα τα παλιά κράτη και επιτέλους αυτά τα τεράστια ελλείμματα που έχουν συσσωρεύσει να τα καλύψουν. Και δεν είναι και καμία δεξιοτεχνία να το αποδείξει κανείς. Τραβάνε τα μαλλιά τους και οι ίδιοι υπάλληλοι και τα στελέχη όταν κοιτάνε τι κάνει το κάθε κράτος μέλος. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα ε, δεν μπορεί να έρθει αυθόρμητα και να ζητήσει οδηγία για τις χωματερές, για τους χιτά έτσι μια οδηγία υψηλή ποιότητα. Κύριε Πρόεδρε, 20 χρόνων αποτυχία δεν χωράνε σε ένα λεπτό. Οι στόχοι μα δεν θα πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμοι, να σκεφτούμε και μακροπρόθεσμου στόχους και την ευελιξία τη ιεραρχία των αποβλήτων. Τι είναι αυτό, αυτό είναι ασθένεια. Είναι Πληγή, γιατί δεν έχουν προτεραιότητε, δεν τις έχουν ορίσει σαφώς και δεν λειτουργούν σωστά αυτά τα πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα και στη Γερμανία παλινοδίες έχουμε και ο ένας μεταθέτει τις ευθύνε στους άλλους. Δεν είναι σαφεί οι κανόνες που έχουμε ψηφίσει, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Πρόεδρε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κατάσταση δεν είναι καλή. Επιτέλους, έχουμε 20 έγγραφα για τις εμβληματικές πρωτοβουλίες. Το flagships αυτά. Ας επιτε... επιτέλους εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε αποφασίσει. Όχι. Ευχαριστώ, θα το πράξουμε ο Βιτόριο Τρία λεπτά αν είναι δυνατόν. Εν συντομία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Επιτροπή για την έκθεση. Ε, θα ήθελα όμως να κάνω και κάποιες προτάσεις για να καταστήσουμε, να, για να καταστήσουμε προφανές στον πολίτη ότι εδώ δεν μιλούμε μόνο για απορρίμματα, αλλά μιλούμε και για πόρους. Επομένως, η διαφοροποιημένη αποκομιδή των απορριμμάτων ε, υπάρχει τεχνολογία για να γίνει και θα πρέπει με επιμέλεια να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις ε, και θα πρέπει το κοινό να αντιληφθεί αυτήν την ε, διαφοροποιημένη αποκομιδή των ε, απορριμμάτων ως έναν τρόπο μείωσης ε, των απορριμμάτων και θα πρέπει να καταστήσουμε κατανοητή την ιδέα ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο τα απορρίμματα και τα απόβλητα αξιολογούνται σωστά και αξιοποιούνται ε, με βάση τη στρατηγική που έχουμε υιοθετήσει. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Chris Θα επαναλάβω λίγο πολύ όσα είπε ο Καρλ Χάιντς Φλόρεντς. Είναι εμβαλωματική η εφαρμογή της νομοθεσίας. Υπάρχουν ορισμένα καλά παραδείγματα και άλλα τα οποία είναι πραγματικά άθλια. Πρόσφατο παράδειγμα, η Ιταλία που δείχνει πόσο άσχημα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Το 2009 η Κομισιόν εξήταζε έγγραφα που συνιστούσαν και πρότειναν την ιδέα ενός οργανισμού εφαρμογής της νομοθεσίας για τα απόβλητα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της δημιουργίας νέων οργανισμών, αλλά τα επιχειρήματα που είχαν προβληθεί με το έγγραφο εκείνο ήταν αρκετά πιστικά. Και δοθήσεις και της δυσκολίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να, προ, να προωθεί συνοδευτικά μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας, ίσως κάποιος τέτοιος οργανισμός να μπορούσε να επιφέρει κάποια διαφορά. Γιατί δεν προωθήθηκε τελικά αυτή η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή γνωρίζει ότι θα είναι θυελώδης η αντίδραση και σημαντική αντίσταση του Συμβουλίου. Και γι' αυτό απέσχει από το να από του να προωθήσει την ιδέα αυτή. Αναμένω την απάντησή σας. Η Χίπνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πόσο δύσκολο είναι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Συχνά οι χώρες μέλη δεν κατανοούν ότι η παραγωγή αποβλήτων και απορριμμάτων είναι τμήμα της οικονομίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραγάγει και ανάπτυξη. Δεν είναι απαραίτητο τα απορρίμματα να είναι βάρος, μπορεί να είναι και κερδοφόρα. Μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη ολόκληρων περιφερειών. Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να γίνουν επενδύσεις στην διαχείριση των αποβλήτων ή απορριμμάτων. Για παράδειγμα, η δημιουργία κέντρων καύσεως ή των περιφημών χιτά, όπου δεν χωράνε πλέον. Έχει, περάσει πια η εποχή των ε, χιτά, των χώρων ε, υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Και ο καθένας εν τέλει πετάει τα σκουπίδια του και όπου θέλει. Η έκθεση αυτή μας λέει, μας δείχνει ότι δεν εφαρμόζουμε την νομοθεσία που ίδιοι έχουμε ψηφίσει. Οι χώρες μέλη ίσως έχουν μεταφέρει την νομοθεσία στα δικιά τους, αλλά δεν την επιβάλλουν. Δεν επιβάλλουν σεβασμό της νομοθεσίας αυτής. Έχουμε ωστόσο δεσμευτικούς κανόνες, αλλά στα χαρτιά. Και συχνά οι χώρες μέλη δεν πράττουν όσα θα έπρεπε. Υπάρχει μέγας κίνδυνος που ήδη διαφαίνεται να δούμε δηλαδή τα απορρίμματα να μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Όπου υπάρχουν χώρες που έχουν παραθυράκια στους νόμους τους, αυτό οδηγεί σε διακίνηση απορριμμάτων μεταξύ χωρών. Αυτό είναι επικίνδυνο. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πραγματικός έλεγχος για το τι συμβαίνει οι χώρες μέλη πρέπει, οφείλουν να ελέγχουν τη διαχείριση των απορριμμάτων και αυτή η διαχείριση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ακόμα ορισμένες, υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις όπως είδατε. Παρακαλώ να μας δώσετε μια απάντηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω για την υποστήριξη που προσφέρει ο κύριος Φλόρεντς στο έργο που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασφαλώς οι προτεραιότητες κατευθύνονται προς την εφαρμογή, αλλά συμφωνώ με, την, με τον κύριο Φλόρενς ότι ο ρυθμός της εφαρμογής και οι διαφορές μεταξύ χωρών είναι πολύ διαφορετικές, είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές δηλαδή. Κάνουμε ωστόσο εμείς εκδηλώσεις για ανταλλαγή πληροφοριών και στις χώρες μέλη και μάλιστα ειδικά πέρυσι για να επιτρέψουμε στις χώρες εκείνες μέλη που εφαρμόζουν και επιτυγχάνουν από τις στρατηγικές τους καλά αποτελέσματα να μπορέσουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους αυτές με άλλες μεταξύ αυτών και των λεγόμενων responsibility schemes και για την για την βολή τελών ε, συλλογής των απορριμμάτων κλπ. Βέβαια, υπάρχουν και καθυστερήσεις στις χώρες μέλη ό,τι αφορά την μεταφορά στα εθνικά τους δίκαια των ε, ε, οδηγιών. Υπενθυμίζω την οδηγία πλαίσιο, όπου η προθεσμία για την μεταφορά ήταν το τέλος του έτους, δηλαδή Δεκέμβριος 2010. Μέχρι τώρα μόνο πέντε χώρες μέλη έχουν περάσει την νομοθεσία αυτή και οχτώ εν μέρη μόνο. Παρόλα αυτά και βεβαίως κάνουμε ε, διαβήματα προς τις χώρες μέλη, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις στην μεταφορά και θα πρέπει να κινηθούν κάποιες διαδικασίες παραβιάσεως. Απαντώντας στα σχόλια ή έστω ως αντίδραση στα σχόλια του κ. Πρόντι, θα πω ότι κάνουμε πολλά πράγματα για να επιτύχουμε την αλλαγή της νοοτροπίας των χωρών μελών σε ό,τι αφορά την θεώρηση των απορριμμάτων ως κάτι που δεν είναι απαραίτητα βάρος αλλά μπορεί να είναι και πόρος και εν προκειμένου πρέπει να τονίσω ότι για πρώτη φορά μπορέσαμε να υιοθετήσουμε κριτήρια για ε, ρινίσματα αλουμινίου, αλουμινίου και άλλων μετάλλων και έχει γίνει και η διαδικασία επιτροπολογίας, τέλειωσε την προηγούμενη εβδομάδα, διότι αυτά τα απορρίμματα είναι σημαντικής αξίας και στρατηγικής χρησιμότητας. Και ε, λοιπόν εγκρίθηκαν τα μέτρα αυτά. Τώρα, θα έχουμε κανόνες που επιτρέπουν να φύγουν από τον έλεγχο των απορριμμάτων τα υλικά αυτά και να χρησιμοποιηθούν πλήρως ως δευτερεύουσες πρώτες ύλες. Για το σχόλιο του κυρίου Ντέιβις για την δημιουργία του Οργανισμού Διαχειρίσεως Απορριμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα αυτή, το ενδιαφέρον της δηλαδή για την ίδρυση αυτού του οργανισμού. Έχουμε διεξαγάγει μια ανάλυση και μια πρώτη μελέτη σκοπιμότητας για τον οργανισμό που έγινε το 2009 και στις αρχές του 2010 δείξαμε τα θετικά αποτελέσματα και εξακολουθούμε να αναλύουμε την σκοπιμότητα μια νέα τέτοια δομή. Διότι γνωρίζουμε ότι η πρότασή μα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ στέρεα. Να αντέχει δηλαδή και στην ανάλυση από οποιαδήποτε πλευρά. Και όσων δηλαδή ενδεχομένω θα ήταν αντίθετη. Για την ώρα αναλύουμε ποσοτικά τα οικονομικά ευεργετήματα των ζημιών που έχουμε από αυτή την ε, ε, ελλείψη στην εφαρμογή και κάνουμε, κόστος, και κάνουμε ανάλυση κόστους ωφέλους. Αναμένουμε αποτελέσματα το φθινόπωρο του 2011 και όπως είπε ο ίδιος ο Επίτροπος πρόσφατα, βασισμένοι στις αναλύσεις αυτές, τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών, θα υποβάλουμε φέτος ακόμη πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι επεισόδια όπως αυτό το πρόσφατο της Ουγγαρίας δείχνουν ότι πρέπει να προωθήσουμε νέες πρωτοβουλίες που να εξασφαλίζουν καλύτερη εφαρμογή των νομοθεσιών, κυρίως όπου η διαχείριση των απορριμμάτων ενδέχεται να επιφέρει κινδύνους στο περιβάλλον ή στην ε, ανθρώπινη υγεία ή να έχει διαμεθοριακές επιπτώσεις. Και μιας και είπα διαμεθοριακές, να σας πω κάποια πληροφορία για τις μετακινήσεις απορριμμάτων. Σημαντικό μέρος αυτό της, της ερώτησης της κυρίας Χίπνερ. Εν προκειμένου η έκθεση δείχνει ότι επιθεωρήσεις φορτίων διεξάγονται, αλλά έχουν και εκεί ελλείψει οι χώρε μέλη. Ω Κομισιόν έχουμε λάβει ορισμένα μέτρα για την βελτίωση των σχετικών κανονισμών, ανταλλαγή πληροφοριών, εκστρατείες συνειδητοποίηση, ε, κατευθύνσει, επίση για τι ανταλλαγέ πληροφοριών για τις, ε, στο εθνικό επίπεδο δηλαδή για τις μετακινήσεις ή τις ε, μετακίνηση φορτίων απορριμμάτων και ειδικά για τα, μέσα ναι, στα πλαίσια της οδηγίας ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών, ώστε αυτά να γίνουν δεσμευτικά. Πρόσθετες guidelines για να γίνει διάκριση μεταξύ επικίνδυνων και μη επικίνδυνων φορτίων και εργαζόμαστε ώστε να κάνουμε πιο εύκολη την εφαρμογή της Και η τελευταία και η πιο σημαντική ίσως πρωτοβουλία στο προκείμενο πλαίσιο είναι ότι στην έκθεση των ε, W3E ε έχουμε μεταφέρει και το βάρος της απόδειξης ότι δηλαδή πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι απορρίμματα. Εν πάση περιπτώσει είναι σαφές ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επιτελούμε πρόοδο και ελπίζω να μπορώ να προσέρχομαι περιοδικά και να σας ε, ενημερώνω για την πρόοδο αυτή. Μάλιστα το θέμα ήταν σημαντικό, λέει ο πρόεδρος Γιώ Θα παραμείνουμε, θα καυτηριάζουμε ξανά και ξανά την έλλειψη εφαρμογής. Θα πάμε με αντιπροσωπεία και σε μια περιφέρεια που είναι πραγματικά πολύ προβληματική, στην καμπάνια της Ιταλίας, Καλαβρία, όπου σημειώνονται σημαντικές ελλείψεις. Θα συνεχίσουμε γιατί στις 4 θα έλθει ο Επίτροπος Έτιγκερ και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εξακολουθούμε να συνομιλούμε με την κυρία Μπλάνκο για την εξαίρεση της απαγόρευσης χρήσεως καδμίου σε φορητές ηλεκτρικές στήλες ορισμένων ε, ασυρμάτων ηλεκτρικών εργαλείων. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη επ' να σας θυμίσω το πλαίσιο. Έχουμε τη νέα οδηγία που εγκρίναμε για τις μπαταρίες το 2006 για να βελτιωθεί η επίδοση συσσωρευτών και μπαταριών προς το περιβάλλον. Αυτό αφορά την κυκλοφορία στην αγορά ε, φορητών ηλεκτρικών στυλών και συσσωρευτών που περιέχουν ε, ε, υδράργυρο και κάδμιο και υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αυτό σε ό,τι αφορά τις συσσωρευτές και τις μπαταρίες ε, σε συσκευές ασύρματες. Είμαστε υποχρεωμένοι να το αναφέρουμε αυτό το θέμα της εξαίρεσης, ε, όπερ και γέννητο το 2010 ε, το Δεκέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολλές μελέτες και εκτιμήσεις αντικτύπου, βαθύτατη ανάλυση και πρέπει να σας πούμε ότι δεν έχουμε στα στοιχεία και επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε την άρση της εξαίρεσης. Είναι σαφές ότι το λίθιο, ε, το νικέλιο και ο σίδηρος και ε, κάποια κράματα τους μπορεί να είναι ε, πιστικές εναλλακτικές ε, λύσεις και υλικά, αλλά έχουν και μειονεκτήματα σε ό,τι αφορά χαμηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης και χαμηλότερη διάρκεια ζωής. Αν καταργηθεί η εξαίρεση, μπορεί να υπάρξει κάποιο πλεονέκτημα ή κάποια ωφέλεια για το περιβάλλον, αλλά δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε κατά πόσο αυτή θα είναι μεγάλη πολύ επισφαλής εκτίμηση. Δεν έχουμε ακόμα αποδείξει ότι το όφελος θα ήταν μεγαλύτερο από το κόστος. Και βασικό συμπέρασμα λοιπόν στην έκθεση κύριε Πρόεδρε στο παρόν στάδιο είναι ότι δεν θεωρούμε σκόπιμο να καταργηθεί η εξαίρεση ε, για το κάθμιο σε φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. Ωστόσο δεν τελειώνει εδώ η υπόθεση. Θα ε, συνεχίσουμε το έργο μας και θα κάνουμε μια εκτίμηση συγκριτική του κύκλου ζωής των υλικών αυτών. Διαβουλευτήκαμε με τους ενδιαφερομένους ε, πέρυσι το Μάρτιο μέχρι και το Μάιο με βάση όλες τις αναλύσεις που κάναμε και όλα τα στοιχεία γιατί πρέπει να σας πω ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν και θεωρούν κατά πλειοψηφία ότι χρειάζεται μια σύγκριση του κύκλου ζωής των διαφόρων τεχνολογικών δυνατοτήτων που έχουμε σήμερα. Είναι τρεις τεχνολογίες, νικέλιο καύμιο, νικέλιο μεταλλικό υβρίδιο και μία τρίτη δυνατότητα και δεν έχουν συγκριθεί μεταξύ τους αυτά τα τρία. Πέρσι τον Οκτώβριο αποφασίσαμε να προβούμε σε αυτή τη συγκριτική μελέτη. Παραγγείλαμε μελέτη η οποία ολοκληρώνεται φέτος τον Οκτώβριο. Τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο ε, θα έχουμε μια ενδιάμεση εκτίμηση, θα έχουμε ένα προσωρινό αποτέλεσμα και θα μπορέσουμε να αρχίσουμε τη σχετική συζήτηση και πάλι θα έχουμε την ευκαιρία να συμβουλευτούμε τους ενδιαφερομένους του κλάδου γιατί γίνεται βαθύτατη ανάλυση, πολύ μεθοδική και μελέτη και συγκριτική όπως σας είπα των τριών τεχνολογιών αν ε, αποδείξει ότι από πλευράς διάρκειας του βίου αυτών των υλικών μπορούμε να βρούμε ε, εναλλακτική πρόταση στην τεχνολογία του καθμίου που θα είναι γενικά εποφελής καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του υλικού, τότε θα σας κάνουμε νέα πρόταση στους συνομοθέτες πιθανότατα αρχές του 2012. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you, Blanco. Chris Davis. Ευχαριστώ, Chris Davis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι ωφέλειες ε, δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερες από το κόστος. Όταν είδα αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη θεώρησα ότι εγγράφει και διότι οι εναλλακτικές λύσεις προς το κάθμιο δεν ήταν αρκετά ε, ποιοτικέ για να βεβαιωθούμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν συσκευέ. Ε, όχι, το site της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σελίδα λέει ότι παραμένουν ε, όμως εναλλακτικέ ε, λύσεις ενισχύ, μπορεί να είναι τοξικές, αλλά είναι λιγότερο τοξικές ή λιγότερο επικίνδυνες από το κάδμιο. Θα ήθελα εγώ να αντιστρέψω το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάπου θα πρέπει να ισχύει και η αρχή της προφύλαξης και κάπου να το γράψει και σε ένα χαρτί Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να αποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το κόστος άρσης της εξαίρεσης είναι μεγαλύτερο από τις ωφέλειες. At the moment the Commission cannot... Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αποφανθεί για το ύψος του κόστους, αν θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το όφελος, γιατί δεν έχουμε ανάλυση ενός πλήρους κύκλου ζωής του υλικού. Λέτε για τα στοιχεία της ε, ιστοσελίδας, δεν είναι μόνο η χρήση, είναι και όλη η παρασκευή, η παραγωγή, η κατασκευή από την αρχή της φάσης και η συνέχεια η διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση τέτοιων ε, συσσωρευτών και μπαταριών. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ε, όσον αφορά την παραγωγή αποβλήτων, έχουμε ενδείξει ότι η αντικατάσταση ε, ε, βαταριών που περιέχουν κάδμιο με μετάλλευμα νικελίου ή κράμα νικελίου ε, σιδήρου θα αυξήσουν την παραγωγή αποβλήτων. Οπότε αυτό αντισταθμίζει λίγο το όφελος της αντικατάστασης του καδμίου. Δεν είμαστε σήμερα όμως σε θέση να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. χωρίς να είναι επίμαχο. αν Διαφυσβήτητο. Γι' αυτό σας είπα ότι θα συγκρίνουμε τρεις τεχνολογίες μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή, κύριε Ντέβις, λυπάμαι και φοβούμαι ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω προς καμία από τις δύο κατευθύνσεις. Γι' αυτό η πιο ειλικρινής ε, απάντηση από πλευρά μα είναι να πούμε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε. Ε, πιέσεις δεχόμαστε κατέρωθεν και ισχυρέ και θα πρέπει να έχουμε και διάστα στοιχεία για να μπορέσουμε να λάβουμε ε, αποφάσεις σε γερό επιστημονικό έδαφος. Σήμερα δεν έχουμε αυτή την κατάσταση. Ελπίζω πάρα πολύ όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση κύκλου ζωής των τριών τεχνολογιών να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα αδιάστα. Ευχαριστώ. Yeah, thank Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Λάινεν. Δεν βλέπω άλλους συναδέλφους να επιθυμούν να θέσουν ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Άρα φαίνεται πως συζητήθηκε και εξετάστηκε εξαντλητικά από στιγμή σε στιγμή αναμένουμε τον Επίτροπο. Επιτρέψτε μου να ανακοινώσω λίγα πράγματα που ήδη είναι από την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Μπανκόκ έγινε η πρώτη διάσκεψη προστασίας του περιβάλλοντος προπαρασκευαστικά για το Durban και όπως ακούω από την Κομισιόν, όπως πάντα, επί της ουσίας δεν σημειώθηκαν σχεδόν καθόλου πρόοδοι. Το καυτό θέμα είναι η συνέχιση της ισχύω του πρωτοκόλου του Κιώτο και το χάσμα μεταξύ βιομηχανικών χωρών και αναπτυσσόμενων χωρών είναι μεγάλο ε, σε αυτό το θέμα του Κιώτο. Δηλαδή η επόμενη συνάντηση προβλέπεται τον Ιούνιο στην Βόνη όπου θα συζητηθούν συγκεκριμένες υποχρώσεις μειώσεων. Τώρα για τη χρηματοδότηση της προστασίας του κλίματος υπέβαλε την Παρασκευή η έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κινητοποίηση πόρων ε, για την ε, προστασία του κλίματος ε, αυτά τα περίφημα 100 δισεκατομμύρια δολάρια που θα πρέπει να ξεβρεθούν μέχρι το 2020 και νομίζω θα μας απασχολήσουν ακόμα πολλές φορές. Την επόμενη εβδομάδα, η επόμενη εβδομάδα μάλλον είναι η λεγόμενη Sustainability Week. Έχουμε και την πράσινη εβδομάδα κάποια στιγμή τον, εβδομάδα κάποια στιγμή τον Μάιο. Την επόμενη λοιπόν εβδομάδα είναι η εβδομάδα της αηφορίας. Εδώ ο κύριος Έτιγκερ, ο επίτροπος κύριος Έτιγκερ, έχει κάνει μια ανακοίνωση για ευφυείς μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια θα μας τα πει και ο ίδιος σε λίγο και μπορούμε να τον ρωτήσουμε για τα θέματα αυτά προσωπικά. Την Τετάρτη της τρέχουσας εβδομάδας έχουμε την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενέργεια, η οποία φαίνεται ότι θα γίνει πιο ακριβή και αυτό ε, προκαλεί μεγάλο θόρυβο, ιδίως στη Γερμανία, στον τύπο. Στις 4 Πέμπτου η Κομισιόν θα υποβάλει τη νέα της στρατηγική βιοπικιλότητας. Αυτές λοιπόν ήταν σύντομα οι ανακοινώσεις προς τις και τους συναδέλφους. Ο κύριος Φλόρεντς έχει μια παρατήρηση για την συζήτηση για τα απορρίμματα. Ευχαριστώ που δέχεστε να λάβω το λόγο κύριε Πρόεδρε. Προηγουμένως λίγο πολύ συμφωνήσαμε και το θέμα είναι διαδικαστικό. Σε τέτοιες συζητήσεις όπου τα είπε καθαρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να προσκαλέσουμε τις κυρίες και κυρίους πρέσβεις του περιβάλλοντος για να πούμε δυο ξεκάθαρα λόγια μαζί τους. Είμαι βέβαιος, απαντά ο Πρόεδρος, ότι το Συμβούλιο Υπουργών όχι μόνο είναι παρόν, αλλά και ακούει προσεκτικά. Και το μήνυμα σίγουρα, η πιθανότατα, έχει περάσει. Αυτό που με εκπλήσει λίγο είναι ότι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν είναι κανένα μέλος της ομάδας των Πρασίνων. Άλλες πολιτικές ομάδες είναι εδώ. Φαίνεται πως έχουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα να κάνουν σήμερα. Θα κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο διάλειμμα και μόλις έρθει ο Γκίντερ Έτινια θα έχουμε σίγουρα ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε μαζί του. So, liebe und Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να προχωρήσουμε στο θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης. Με χαρά καλωσορίζω στην Επιτροπή μας τον Επίτροπο κύριο Έτινγκερ. Κύριε Έτινγκερ, δύο φορές έχετε έρθει να μας δείτε κάθε φορά που συνέβαινε κάποια καταστροφή την προηγούμενη χρονιά στις 5 Εβδόμου μετά από την έκρηξη της πλατφόρμας στον κόλπο του Μεξικού και τώρα πρόσφατα μετά από τα συμβάντα στην Ιαπωνία. Η σημερινή συνεδρίαση δεν είναι συνεδρία καταστροφής, συνεδρίαση καταστροφής, το πω έτσι, αλλά είναι τακτική συνεδρίαση στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου που διεξάγεται μεταξύ με, ε, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια των σχετικών ρυθμίσεων. Θα ακούσουμε τον σχεδιασμό σας για την ενεργειακή πολιτική που είναι το μέγα θέμα που απασχολεί βεβαίως πρωτίστως την Επιτροπή Βιομηχανίας αλλά και την δική μας Επιτροπή για πολλούς αποχρόντες λόγους. Οι συνάδελφοί μου ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το τι έχετε στα χαρτιά για φέτος αλλά και για του χρόνου. Γνωρίζω ότι μετά το Στρασβούργο έρχεστε μετά από επίσκεψη μεγάλης πλατφόρμας της Βίντε στην Βόρεια Θάλασσα που σίγουρα θα ήταν ε, σημαντική ε, επίσκεψη. Πρόκειται για ε, αιωλική ενέργεια που συλλέγεται εκεί και που ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και με χαμηλό κόστος για όλη την Ευρώπη. Ο κύριος Έτιγερ, αγαπητέ κύριε Λάινεν, κυρίες και κύριοι, στις σύντομες προκαταρκτικές μου παρατηρήσεις θα περιοριστώ σε τρία θέματα στις δραστηριότητες offshore για το αέριο και το πετρέλαιο, δεύτερον πυρηνική ασφάλεια και μετά το εργοστάσιο Φουκουσίμα και τρίτο αποδοτικότητα της ενέργειας και τι πράττουμε για να προχωρήσουμε για να διατηρήσουμε την πρωτοπορία μας στην αποδοτικότητα της ενέργειας. Επίσης θα ήθελα σήμερα στην συζήτηση να έλθω και στην ημερήσια διάταξη που μας απασχολεί για να τη συζητήσω μαζί σας, αφενός δηλαδή τους γενικούς στόχους 2020, δεύτερο την ενιαία αγορά και την ολοκλήρωσή της, τρίτο το θέμα υποδομές ενέργειας και κυρίως ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου. Τέταρτο, τις προπαρακευαστικές μας ενέργειες για την εξωτερική πολιτική ενέργειας και τον διεθνή ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέμπτο, την από Μαΐου σε μακροπρόθεσμη αποστολή για, την, για την, με χρονικό ορίζοντα 2050 πλέον που θα συζητηθεί και με τα άλλα κοινοβούλια. Πρώτα, στην γενική μας διεύθυνση κάνουμε ε, αξιολόγηση των επιπτώσεων μετά από την ανακοίνωσή μας του περασμένου Οκτωβρίου. Έχουμε αρχίσει και μια ε, δημόσια ακρόαση. Συνεχίζουμε την διαβούλευση με τους Ευρωπαίους πολίτες σε όλα τα θέματα offshore. Και αυτό μέχρι τις 11 Μαΐου. Για θέματα ασφαλείας δηλαδή των ε, παράκτιων ε, ε, εκμεταλλεύσεων. Έχουμε διάλογο με μη κρατικού οργανισμούς, με επιχειρήσεις και βεβαίως η βιομηχανία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Θα υποβάλουν προτάσεις και για μέτρα για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Εδώ ασκούμε πίεση και αναμένουμε συγκεκριμένες προσφορές από πλευρά της βιομηχανίας μέχρι το καλοκαίρι φέτος. Σύμφωνα και με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σας για την ασφάλεια των ε, πηγών offshore, θα φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ισχύσουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι πρακτικές οι οποίες έχουν μέχρι τώρα αποδείξει την αξία τους. Για παράδειγμα και άλλες και από Νορβηγία. Υπάρχουν κενά ε, στην νομοθεσία και ιδίω ε, στην οδηγία της ε, ευθύνη για ζημίε στο περιβάλλον, τα οποία και να θέλουμε να κλείσουμε, αλλά βέβαια πρέπει να γίνουν και πιο ευνόητοι οι κανόνες. Άρα χρειάζεται κατάρτιση και περαιτέρω κατάρτιση των εργαζομένων, μεγάλη σημασία σε αυτό. Οι ίδιες οι αρχές πρέπει να συμβάλλουν ώστε οι ελάχιστες απαιτήσει που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο κατανοητές και να εφαρμόζονται. Όσο πιο ενιαίας μορφής είναι οι απαιτήσει αυτές και όσο πιο εύκολο να εφαρμοστούν, τόσο μεγαλύτερη σαφήνεια μπορεί να επιτευχθεί. Και ασφάλεια επομένω. Θέλουμε να φροντίσουμε επίση σε ό,τι αφορά τι διατάξει για την χορήγηση εγκρίσεων. Αυτέ να συγκλίνουν περισσότερο, δηλαδή να μην μεταφέρονται οι αρμοδιότητε, αλλά να υπάρχουν κοινέ απαιτήσει και τεχνικέ και περιβαλλοντικέ και ε, οικονομικού χαρακτήρα. Κάθε επιχείρηση η οποία ε, ζητεί μια χορήγηση έγκριση να υπάγεται ακριβώ στι ίδιε απαιτήσει, όπου, οπουδήποτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αυτό. Εγώ βρίσκω ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό εδώ για την βελτίωση τη ανταλλαγή πληροφοριών και την διαφάνεια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κεντρικό, ένας συνομιλητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση ατυχημάτων σε πλωτές δεξαμενές και ούτω καθεξής. Εξάλλου θέλουμε όλες οι ρυθμιστικές αρχές των offshore να προσέλθουν σε μια τράπεζα για να συζητήσουν κοινέ, σε μια τράπεζα για να συζητήσουν κοινέ προδιαγραφές και να τις προωθήσουν. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν τέτοιες δομές ευρωπαϊκών διαστάσεων. Τα συμφερόντά μας λοιπόν, αλλά και τα ενδιαφέροντά μας και πέραν των συνόρων μας, διότι οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην Μεσόγειο μας δείχνουν ότι η ασφάλεια και των γειτονικών μας περιοχών οφείλει να ελκύσει την προσοχή μας. Για παράδειγμα, Λιβύη. Γι' αυτό και μετά από τις ανατρεπτικές αυτές εξελίξεις θέλουμε μαζί με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενέργειας να μπορέσουν να εξαγάγουν κιόλας τις απαιτήσεις αυτές τις οποίες ανέφερα προηγουμένως και σε άλλες περιοχές του κόσμου οι οποίες συνδέονται ή είναι γειτονικέ μαζί μας, όπως ο χώρος της Μεσογείου. Ο σχεδιασμός μας μετά από τις ακροάσεις και διαβουλεύσεις προβλέπει πριν από το καλοκαίρι να καταθέσουμε σχετική πρόταση και αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την δική σας θέση, θέση καθώς και πρόκειται να συνεργαστώ μαζί σας, καθώς και με το Συμβούλιο Υπουργών και πριν από το καλοκαίρι και μετά. Δεύτερο, πυρηνικά θέματα τώρα. Γνωρίζετε ότι έχουμε προτείνει και έχουμε αρχίσει δοκιμασία αντοχής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φάνηκε μετά από τα ε, φοβερά συμβάντα του Φουκουσίμα ότι ανεξαρτήτως θέσεως μπορεί να έχει κανείς για την πυρηνική ενέργεια και ότι υπάρχει μία κοινή απέτηση της ύψης της δυνατής ασφάλειας υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό και κάναμε την πρόταση δοκιμασιών αντοχής που εγκρίθηκε από το Συμβουλίο Υπουργών και έδωσε αυτό την σχετική εντολή. με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μας ήταν σημαντικό για να διατηρηθεί η ενότητα των δοκιμασιών αντοχής να μην γίνουν μονάχα εντό εισαγωγικών από τις εθνικές εποπτικές αρχές αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με διασταυρούμενους ελέγχους ώστε να γίνει κατά το δυνατόν κοινή η διαδικασία, κοινή η προσπάθεια αυτή των δοκιμασιών αντοχής και η απόφαση του Συμβουλίου ε, κινήθηκε προς την διακατεύθυνση. Μαζί με την INSREC λοιπόν κάνουμε τώρα ε, εξέταση των κριτηρίων, των κέντρων βάρους, της διαδικασίας και θέλουμε κοινή εφαρμογή για να δείξουμε καθαρά και τον διαμεθοριακό, τη διαμεθοριακή υπερσυνοριακή φύση ενδεχόμενων πυρηνικών ατυχημάτων με κοινά κριτήρια καθώς και τις λεγόμενες peer reviews που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Και αυτά υπό πλήρη διαφάνεια. Σας υποσχέθηκα ήδη πλήρη διαφάνεια και για την εξέταση των κοινών κριτηρίων πριν και για την εκτέλεση των δοκιμασίων αντοχής, αλλά και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Απόλυτη διαφάνεια απέναντι στο Κοινοβούλιο, μη κρατικού οργανισμού και ούτω καθεξής. Με την έννοια αυτή, τα αποτελέσματα των δοκιμασίων αντοχής θα τα εξετάσουμε μαζί με το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα τα αξιολογήσουμε και θα τα περιλάβουμε σε έκθεση την οποία θα σας υποβάλλουμε που μπορεί να είναι σημαντική για την περαιτέρω εργασία σας. Έχουμε προβλέψει και μία συνάντηση μετά από το Πάσχα με, τους, με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους stakeholder και 12 και 13 Μαΐου να εγκρίνουμε τα κριτήρια στην ετήσια συνεδρίαση της Ινσρεκ θα συναντηθώ μαζί σας ή με τους συντονιστές σας τις δύο πρώτες εβδομάδες του Μαΐου, επομένως πριν από αυτή την ετήσια σύνοδο της Ίνσρεκ, ώστε να διεξαγάγω περαιτέρω συζητήσεις μαζί σας για να ακούσω τις ενδεχόμενες επικοδομητικές σας προτάσεις. Το ίδιο προσφορά διαλόγου και προς τους μη κρατικούς οργανισμούς που εργάζονται στο τομέα αυτό, στον κλάδο αυτό. Η αξιολόγηση του κινδύνου αρχίζει πρώτα σε βάση μιας ε, ενιαίας μεθόδου από τους ίδιους τους φορείς της βιομηχανίας. Και αυτό θα αποτελέσει και τη βάση για τις peer reviews που είναι απαραίτητες, είναι κρίσιμη σημασία. Θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις και, ε, και άποψη των εποπτικών αρχών, αλλά και οι peer reviews που όπως είπα είναι πάρα πολύ σημαντικές για να υπάρξει μια νέα ευρωπαϊκή εποπτεία και για να εξασφαλιστεί ώστε στις διάφορες επιμέρους χώρες μέλη να γίνεται η προσέγγιση της αξιολογήσης με τον ίδιο τρόπο. Εγκαταλείπουμε έτσι την μέχρι τώρα πρακτική του ελέγχου εντός της επιχείρησης και από τις εθνικές εποπτικές αρχές, για έτσι για πρώτη φορά ερχόμαστε στο ε, ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε διασταυρωμένους ελέγχους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια μέχρι τέλος του 2011. Γνωρίζετε ότι από τον Ιούνιο του 2009 υπάρχει και μια οδηγία, ε, Ευρωπαϊκή Οδηγία Πυρηνικής Ασφάλειας, η οποία βρίσκεται στην φάση μεταφοράς στα εθνικά δίκαια στις ε, χώρες μέλη που θα ε, ισχύσει μέχρι τον Ιούνιο και που προβλέπει μέχρι το 2014 να γίνει αξιολόγηση. Τώρα αυτό προτάσεται και βάζουν μέχρι τέλους του 2011 και για θέματα τυπικά της ε, πυρηνικής εποπτείας και για ουσιαστικά ζητήματα της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας όπου θα κάνουμε πρόταση για την μορφή που θα πρέπει να λάβει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, για την οδηγία δηλαδή, και πώς αυτή θα εμβαθυνθεί. Αυτή η διαδικασία εκ θα, θα γίνει εκ παραλίλου με τις δοκιμασίες αντοχής που θα μας οδηγήσουν σε περαιτέρω ε, εξαγωγή συμπερασμάτων. Αποδίδουμε αξία στο ότι οι ευρωπαϊκές ε, χώρες μέλη θα πρέπει μέχρι τις, των αρχών Ιουλίου να έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία που ανέφερα προηγουμένως για την πυρηνική ασφάλεια καθώς επίσης και για τα απόβλητα, η οποία τώρα υπό το φως των συμβάντων στην Ιαπωνία αποκτά αυξημένη σημασία. Εργαζόμαστε τώρα επί της διαμόρφωσης των ε, stress test, των δοκιμασιών αντοχής για την πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη, αλλά να επεκταθούν αυτές οι βασικές αρχές και σε χώρες εκτός Ευρώπης, ιδίως στην Ουκρανία, με την οποία βρισκόμαστε σε συζήτηση, με την Ρωσική Κοινοπολιτεία, επίση διεξάγουμε διάλογο, την Ελβετία, με την οποία θα αρχίσουν οι συζητήσει την επόμενη εβδομάδα, και την Αρμενία. Πέραν αυτού, θέλουμε να ε, διεξαγάγουμε διάλογο και με χώρες οι οποίες σκέπτονται ή σχεδιάζουν ή προετοιμάζουν την κατασκευή πυρηνικών σταθμών, ιδίω την Τουρκία ή την Λευκορωσία. Θέλουμε δηλαδή ή δυνατόν μια εταιρική σχέση που να υπερβαίνει τα ε, όρια της Ευρώπης. Εν τέλει, τελευταίο θέμα για σήμερα, αποδοτικότητα της ενέργειας. Έχετε λάβει την πρότασή μας. Όλο και μεγαλύτερη γίνεται η σημασία της αποδοτικότητας της ενέργειας. Ακόμα απέχουμε σημαντικά από τους στόχους μας. Ένα κεντρικό θέμα θα είναι ο τομέας των κτηρίων. Μέσα στο νέο μας σχέδιο δράσεως θα προβλέψουμε συγκεκριμένες υποχρεωτικές απαιτήσει για τα δημόσια κτίρια. Δημόσια κτίρια, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κλινικές, ακόμα και παιδικοί σταθμοί, στρατώνες, που εν πάση περιπτώσει συναπαρτίζουν το 12% όλων των κτίριων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θέλουμε αυτό το ποσοστό σταδιακής ανανέωσης ανακαίνησης των κτηρίων που είναι αυτή τη στιγμή στο 1,2-1,5% ανέβει τουλάχιστον στο 3%. 3% είναι ήδη αρκετά δυσχερές. Υπάρχουν φωνές, κυρίως από την πλευρά των αρμοδίων του προϋπολογισμού, που λένε ότι τους φαίνεται υπερβολικά υψηλό το ποσοστό αυτό. Αλλά 3% σημαίνει 33 χρόνια. Υπάρχει όμως ε, και ο χαρακτήρας υποδείγματος των δημοσίων αρχών που δεν πρέπει να λησμονείται. Δηλαδή θα αποτελέσουν και παράδειγμα για τους υπολείπους, για τους πολίτες. Και ιδίως βεβαίω θα πρέπει το καλό παράδειγμα να δώσουν τα κτίρια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Επανέρχομαι στην βιομηχανία. Και στη βιομηχανία η ενεργειακή αποδοτικότητα ε, έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα εξαναγκαστούν με ελέγχους απόδοσης ενέργειας και με τα σχετικά συστήματα και για μικρές και μεσές επιχειρήσεις προβλέπουμε περιορισμένου χαρακτήρα μέτρα. Έχουμε μια στατική δύο σταδίων μέχρι το 2012-2013 σε εθελοντική βάση. Αν δούμε όμως το 2013 ότι δεν επιτυγχάνονται τα 20%, ότι ίσως τα βήματα είναι πολύ μικρά ή διστακτικά, τότε, και το ανακοινώνουμε ήδη σήμερα, από το 2014 και μετά θα προχωρήσουμε σε δεσμευτικές απαιτήσει για τα επόμενα 6-7 χρόνια, για να φτάσουν δηλαδή μέχρι το 2020. Ήδη τούτο τον μήνα θα ε, εκδώσει την ανακοίνωσή της για το λεγόμενο FES δίκτυο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό θα είναι μέρος της πολιτικής μας για την αύξηση της αποδοτικότητα της ενέργειας. Επίσης, για του λεγόμενους ευφυεί e μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι όμως ακόμη επαρκές. Γι' αυτό εξετάζουμε ξανά ολόκληρη την αρχιτεκτονική των λεγόμενων ευφυών e δικτύων από το κέντρο του δικτύου μέχρι και τον τελευταίο μετρητή. Να είναι ένα ανεπτυγμένο τεχνολογικό δίκτυο. Εδώ προβλέπονται εξή τομεί. Πρώτο, ανάπτυξη ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για τους ευφυείς μετρητές. Δεύτερο, εξασφάλιση προστασίας δεδομένων του καταναλωτού, να μην υπάρξει δηλαδή ενδεχόμενο κατάχρησης ε, διαδραστικά των δικαιωμάτων του ε, καταναλωτή. Επίσης, δημιουργία πλαισίου για την χορήγηση κινήτρων για την δημιουργία των ε, ευφυών μετρητών διατάξεις για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστική αγοράς εποφελία του καταναλωτού και συνεχή προώθηση τεχνολογικών συστημάτων, ειδικώ βέβαια για να εξελιχθεί και να προωθηθεί και η έρευνα στους τομείς αυτούς. Προετοιμάζουμε και την πρωτοβουλία μας για τις λεγόμενες ευφυείς πόλεις, οι κέντρα και κοινότητες, που εν τέλει εκεί κατοικούν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πολιτών για το θέμα της ε, κατανάλωσης ενέργειας, κινητικότητα και συγκοινωνίες και μαζί με τον ε, συνάδελφό μου επίτροπο κύριο Κάλλας μελετώ ένα πρόγραμμα πρότυπου χαρακτήρα όπου το θέμα της αποδοτικότητας της ενέργειας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά λοιπόν για την ώρα είναι τα τρία βασικά κέντρα ενδιαφέροντός μας και που ε, θα συνεχίσουν να μας απασχολούν σε όλο το 2011. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλα θέματα που ενδιαφέρουν και το κοινό. Με χαρά δεχόμαστε την πρόσκλησή σας πριν την ετήσια συνεδρίαση της ΕΝΣΡΕΚ να συνεννοηθούμε με τους συντονιστές και με τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας να δούμε τα κριτήρια μέτρησης ε, και δοκιμασίας, να μην τα μάθουμε από τις εφημερίδες, θα βρούμε μια ημερομηνία. Ε, οι υπεράκτιες ε, δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου, ε, πήρατε μια επιστολή από την Κύπρο νομίζω για τον τρόπο που θα γίνουν όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί ήδη. Ε, αν στη συνέχεια έχετε να πει τίποτα για ε, τον οδικό χάρτη για την ενέργεια για το 2050 γιατί είναι μεγάλη κύκλη των επενδύσεων την ενέργεια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλες εγκαταστάσεις και πρόκειται για πολλά δισεκατομμύρια, τα οποία θα επενδυθούν προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Οπότε νομίζω θα πρέπει να δοθεί ε, μία κατεύθυνση πορείας να ξέρουμε που βαδίζουμε ε, να μην έχουμε απαρχιωμένε μορφέ ενέργειας το 2050 που τότε θα τι επιθυμούμε. Λοιπόν, ενδιαφέρον ε, προξενήσατε πολλές ε, οι τοποθετήσεις, να κοιτάμε και το ρολόι, δύο λεπτά έκαστος για να προκάνουμε. Ο Χόρστ Σνέλχαρτ πρώτος. Α, Εξεπλάγεν που αρχίζω εγώ πρώτο. Λοιπόν, κύριε πίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχεστε πάντα εδώ και μας παρουσιάζετε τις προθέσεις σα και το πρόγραμμά σας. Θα ήθελα να αρχίσω από την ενεργειακή αποδοτικότητα. Συζητούμε γενικά την οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι χρειάζονται οικονομίες, Ακούμε συνέχεια από τους Δήμους και κοινότητες και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδίκησης ότι το ταμείο είναι μείον. Ιδιαίτερα αυτά τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης, αυτά τα μέτρα κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα. Τώρα δεν ξέρω ποια μέτρα ε, δεν θα εγκαταληφθούν στη θέση τους γιατί κάπου πρέπει να βρεθούν τα χρήματα και κάπου έρχεται σε αντίφαση αυτός ο στόχος αν θέλουμε να τον ε, επιβάλλουμε. Τι θα πούμε, ότι ε, όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν, το χρέος και τα λοιπά, τι ιδέες έχετε για την ε, προσέλκυση πόρων. Κάτι άλλο που με ενδιαφέρει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει μια ανακοίνωση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Εσείς κάνετε τώρα τις δοκιμές αντοχής και μετά από τις δοκιμές αυτές θα κλείσουν ορισμένα πυρηνικά εργοστάσια ή μπορούμε εμείς από την Ευρώπη να το υποδείξουμε έτσι, αν δεν τηρούνται κάποια κριτήρια να ε, κλείσουν τα εργοστάσια αυτά. Και μετά θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Και ποιε θα μπορούσαν να είναι αυτέ, Έχετε κανένα πρόγραμμα, κανένα χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης για το τρίτο, το σύστημα εμπορίας ρήπων. Μόλις το ψηφίσαμε εδώ στην Επιτροπή μας και είπαμε το τρίτο στάδιο από το 2013 είναι εντάξει, ε, προγραμματίζεται, αλλά τώρα βλέπω όλη τη συζήτηση που στρέφεται και άλλες πηγές και ε, όμως και τον άνθρακα και το φυσικό αέριο για να έχουμε εξασφαλισμένη ενεργειακή προμήθεια. Αυτό δεν πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Στο δευτερόλεπτο Κρήτον Αρσένης παρακαλώ. President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε. Αναφέρατε πολλά πράγματα. Θα ήθελα να εγείρω και το ζήτημα της, το πυρηνικό και το θέμα των πυρηνικών επιθέσεων. Υπάρχουν κρυμμένα κόστη στην... Ε, ε, ε, όχι τις πυρηνικές επιθέσεις, αλλά την τιμή της πυρηνικής συνέργειας. Υπάρχουν κρυμμένες τιμές και δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποτιμήσουμε σωστά την κατάσταση αν δεν έχουμε μια λεπληρωμένη εικόνα όλων των κατηγοριών κόστους. Ε, ε, φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα πυρηνικά απόβλητα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους, ε, κινδύν, τον κίνδυνο πυρηνικών ατυχημάτων που όταν συμβαίνουν είναι θέμα διακρατικό. Σκέφτεστε να εγγενιάσετε, να δρομολογήσετε κάποια συζήτηση για τον συντονισμό ή για την επιβολή ενός πυρηνικού φόρου. Ο Κρίς Ντέιβις, Επίτροπε, μου φαίνεται ότι η σημασία της συλλογής και αποθήκευσης άνθρακα έχει υπερτιμηθεί στη θεματολογία. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που το Συμβούλιο ξεκίνησε τους πρώτους στόχους και δρομολόγησε το πρόγραμμα το οποίο θα κατέληγε το 2015. Είναι προφανές ότι δεν θα τα καταφέρουμε μέχρι τότε, η πρόοδος είναι πάρα πολύ αργή και στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας υπάρχουν έξι μεγάλα σχέδια τα οποία υποστηρίζονται από οικονομικά προγράμματα. Μερικά από αυτά όμως δεν έχουν εξελιχθεί και πολύ γρήγορα. Στη Βρετάνια, για παράδειγμα, δεν γίνονται και πολλά. Επίσης, υπάρχει ένας ενθαρρυντικός αριθμός αιτήσεων για, την, ε, για το μηχανισμό στήριξης ε, για τους σπόρους που προέρχονται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Όλα αυτά οφείλονται μόνο σε αυτή την επιτροπή μας. Αν δεν υπήρχε η επιτροπή μας να θέτει τα ζήματα αυτά, τίποτε δεν θα γινόταν, ούτε ένα λεπτό δεν θα δινόταν. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν για να καταστούν πιο επιτακτικά τα θέματα αυτά και ο σημερινός καταμερισμός εργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης του Περιβάλλοντος και της Γενικής Διεύθυνσης της Ενέργειας. Νομίζω ότι η Γενική Διεύθυνση της Ενέργειας θα παίξει ε, πολύ μεγάλο ρόλο. Εάν πρόκειται να έχουμε μια ειδική στρατηγική για τον άνθρακα, τότε σίγουρα η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας θα πρέπει να, να στηρίξει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Ήταν εισηγητής ο ε, για αυτά τα θέματα, γι' αυτό σας ρωτάει. Ε, Μορκουνάιτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, ε, πρόκειται να παρουσιαστεί μια ανακοίνωση για την ασφάλεια της ενέργειας, του εφοδιασμού και τη δημόσια συνεργασία και την κρατική συνεργασία. Ε, το Συμβούλιο των Υπουργών κατέληξε σε πολύ σαφή συμπεράσματα επ' αυτού και μας έδειξε το δρόμο. Το... Μας έδειξε τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτό που θα έχω να πω φυσικά άπτεται τον πυρηνικού ζητήματος. Ε, είπατε πολλά υποσχόμενα πράγματα για τη συνεργασία με τις ε, χώρες που γυτνιάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Ποια είναι η γενική διάθεση ε, στις, τρίτες χώρες, ε, στις τρίτες χώρες, ποια είναι η εντύπωση που αποκομίσετε από τις ε, διμερείς επαφές που έχετε με τις χώρες αυτές και την ανάγκη να εφαρμόζουν αυστηρότερα πρότυπα και κανόνες. Τώρα για την ε, εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, για παράδειγμα, πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από πυρηνική ενέργεια που δεν ανταποκρίνεται στους υψηλούς κανόνες και προδιαγραφές που έχουμε. Ε, θα, τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε απέναντι σε τρίτες χώρες οι οποίες ε, δεν τηρούν τις διεθνείς συμφωνίες για τα πιο αυστηρά ε, πρότυπα. Μήπως προβλέπετε κάποιος μηχανισμός ώστε να μην μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν τιμούν τις υποχρεώσεις τους. Ε, έχουμε και λιθουανική ε, καμπίνα. Θα μπορούσατε να ε, είχατε μιλήσει τη γλώσσα σας. Ο Ζιλ Περνιό. Ευχαριστώ, Επίτροπε. μου αποκόμισα μια πάρα πολύ ευνοϊκή εντύπωση από εσάς, από την τελευταία ακρόαση εδώ, για, για την για το σώμα των εθελοντών που θέλετε να αναπτύξετε για την αντιμετώπιση ε, καταστροφών. Ε, η Επιτροπή θέλει να δει πώς θα γίνει η προώθηση της ε, ενεργειακής ατζέντα στο μέλλον. Πώς θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την ενεργειακή στρατηγική μας από εδώ μέχρι το 2050. Σήμερα είναι λίγο εξασθενημένα τα πράγματα. Έχω την εντύπωση αποκονίζω από, τον, ε, ε, την ομιλία σας ότι δεν δεν υπάρχει αρκετή πεποίθηση πίσω από την ενεργειακή πολιτική. Εσείς μεν εκφράζετε κάποια ισχυρή βούληση ε, και μιλάτε για αυτά τα, αυτές τις δοκιμασίες αντοχής, οι οποίες πρέπει να διεκπεραιωθούν με αντικειμενικότητα και απέναντι στα κράτη-μέλη και απέναντι στην βιομηχανία. Ε, δεν ξέρω τι είδους αντιστάσεις συναντάτε από τα κράτη-μέλη. Από την άλλη, για την κατάρτιση της κοινοτικής στρατηγικής, ε, σας παρακολούθησα μαζί με τον πρόεδρο Μπιζέκ και τον Ζακ ε, Ντελόρ ποια θα, ποιος είναι αυτός ο δρόμος μιας ενεργειακής ε, ευρωπαϊκής πολιτικής. Όταν βλέπουμε τι συμβαίνει στον πυρηνικό τομέα, υπάρχει, νομίζω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τις αναλλακτικές ε, πηγές ενέργειας. Το είπατε άλλωστε κι εσείς. Εσείς ε, Ποια γνώμη έχετε για την αυξανόμενη βούληση ορισμένων μερίδων του πληθυσμού να εγκαταλειφθεί η πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι πρέπει να αλλάξουμε την οπτική μας για το 2050. Θα πρέπει να αποκτήσουμε σωστούς στόχους και να τους υποστηρίξουμε με τη σωστή χρηματοδότηση και γενικότερα. Τι γίνεται με τα... Υπάρχει ένας προϋπολογισμός ο οποίος πηγαίνει στον πυρηνικό τομέα και δεν υπάρχει αντίστοιχος προϋπολογισμός που να διοχετεύεται στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση πρόκειται να εργαστείτε εσείς να, να θέσετε το ζήτημα της μεταβολής των στόχων του 2005, της αλλαγής κατεύθυνσης, αλλά όχι μόνο σε επίπεδο ελπίδων και προσδοκιών, σε επίπεδο πραγματιστικό και σε επίπεδο προϋπολογισμών και πόρων. Δεύτερον, Ε, συμφωνώ και εγώ με αυτή τη σύζευξη μεταξύ του τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Ε, αν κατάλαβα σωστά, ε, σκοπεύετε να κάνετε μια πρόταση πριν από το καλοκαίρι. Πού βρισκόμαστε όσο αφορά την υλοποίηση των κοινοτικών νομοθετικών κανόνων. γιατί δεν υλοποιούνται αυτοί οι κανόνες, για παράδειγμα, στις υπεράκτιες πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου. Θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερα. Ε, τι σχέδια έχετε για τον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προτείνω τώρα ο Επίτροπος να απαντήσει στις έξι πρώτες ερωτήσεις και μετά ε, θα γίνουν και πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Παρακαλώ. Κάποιος ρώτησε τι γίνεται ε, με την χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης. Πραγματικά, τα κτίρια και κυρίως τα δημόσια κτίρια ε, χρειάζονται και ιδιωτικούς πόρους και δημόσιους πόρους, έτσι, συγχρηματοδότηση. Ή ας πούμε ένα σπίτι, 140 τετραγωνικά, μια κατοικία της δεκαετίας του 60. Αν ε, γίνει μόνωση παντού, θερμομόνωση και έχω μόνωση από τη στέγη μέχρι ε, το πάτωμα είναι μια υπόθεση που μπορεί να φτάσει από 60, 70 και 80 ε, χιλιάδες ευρώ. 500 ευρώ το τετραγωνικό είναι καλή επένδυση, αλλά όχι για το λογαριασμό της ενέργειας του επομένου έτους. 30 κοντά ετία είναι ο ορίζοντας. Με λιγότερη ενέργεια δηλαδή και ενεργειακό κόστος αποδίδει αυτό και αποσβαίνεται το κόστος. Το ίδιο ισχύει και για τα κρατικά κτίρια, για τα δημόσια κτίρια. Θα πρέπει ε, να έχουμε ένα κονδύλι στους προϋπολογισμούς ε, σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, κρατικό και ευρωπαϊκό. Τι θέλουμε να προσφέρουμε. Τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ε, ταμεία συνοχής και τα περιφερειακά, που μέχρι τώρα όμως σε περιορισμένο βαθμό συμμετείχαν ε, σε αυτή τη δραστηριότητα. Θέλουμε να το επεκτείνουμε στο βαθμό που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν απορροφηθεί 100% οι πόροι αυτοί. τα μεταφορές πιστώσεων από χρήματα που περίσευαν και δεν είχαν εκταμιευθεί και τελικά χανόντουσαν. Δηλαδή, χωρίς περισσότερη χρηματοδότηση και χωρίς οικονομική επιβάρυνση θα μπορούσε ο κοινοτικό προϋπολογισμός να βοηθήσει να απορροφώνται 100% τα κονδύλια αυτά με μεγαλύτερη εστίαση στην ενεργειακή απόδοση ισχύει αυτό για το δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να ε, ε, ε, λειτουργήσουμε σε επίπεδο που δεν φαίνεται. Δηλαδή μην κάνουμε έργα ωραία βιτρίνας με κοσμητική επέμβαση, δεν θα έχουμε να βάφουμε προσώψεις και τα λοιπά. Δεν είναι ένα θέμα πρεστής και έγκλης, είναι μια δουλειά λίγο πιο αόρατη, αλλά πολύ πιο αποδοτική και θα συμμετέχουν και οι αρχές και ε, με αλλαγή ε, της χρηματοδότησης μεταφορά πιστώσεων ε, σε αυτό το τομέα. το εμπόριο ρήπων και πολιτική της βιομηχανίας. Το καλοκαίρι θα φέρουμε στο Κοινοβούλιο πρόταση ε, για το τι θα γίνει με το σύστημα εμπορίας ρήπων από το 2013 και μετά. Ήδη από τώρα γίνεται μεγάλος αγώνας. Ποιος από τη βιομηχανία, σε ποιο κλάδο, ε, χαλιβουργία, χημεία, τσιμεντοβιομηχανία, ε, ποιο κλάδο της βιομηχανίας έχει πιο, πιο κόστος και ποιο πρέπει να πληρώσει και τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Αυτό το σύστημα εμπορίας ε, ρήπων θα πρέπει να το συνεχίσουμε νομίζω. Είναι χρήσιμο ευρωπαϊκό μέσο και σημαντικό και ακόμα και αν δεν μας ακολουθήσουν άλλες περιοχές του κόσμου για ένα παγκόσμιο σύστημα ETS χρειάζεται ακόμα πολύ πυθό, αλλά από το 2013 να το διαμορφώσουμε έτσι το σύστημα ώστε να μην υπάρχει αναγκαστικός λόγος για κανένα κλάδο της βιομηχανίας να σηκώνεται να φεύγει από την Ευρώπη. Διότι η προστασία του κλίματος δεν εξυπηρετεί το να σηκώνεται και φεύγει ένα εργοστάσιο και μπορεί να εκπέμπει 100% εκτός της Ευρώπης χωρίς κόστος και εμείς να χάνουμε και έσοδα και να χάνουμε και θέσεις απασχόλησης. Δεν έχει νόημα αυτό. Είναι μια τρύπα στο νερό. Θα πρέπει να συνεχιστεί το ETS, ε, αλλά με τρόπο ευέλικτο, έτσι ώστε κανένας μεγάλος αξιόλογος εργοδότης να μην χρειάζεται να φεύγει από την Ευρώπη. Γιατί η παραγωγή θα συνεχίζεται. Δεν χάνεται, δεν εξαφανίζεται, γίνεται κάπου αλλού. Και για μένα κάθε παραγωγή είναι καλύτερο να γίνεται στην Ευρώπη με τις δικές μας προδιαγραφές για το περιβάλλον και τα δικά μας έσοδα για το περιβάλλον και επιτυχάνονται και περισσότερα πράγματα για το περιβάλλον και διατηρούμε και τις θέσεις που δημιουργούν και αξία και κέρδος και φόρους και έσοδα. Επίσης κάποιος ρώτησε τι αλλαγές θα γίνουν μετά ε, τα τρομακτικά συμβάντα στην ε, Ιαπωνία για τη δική μας ε, ασφάλεια του ανεβοθιασμού της ενέργειας και το δικό μας ενεργειακό μείγμα εντός εισαγωγικό. Εάν κλείσουν μόνο 8 πυρηνικά εργοστάσια στη Γερμανία, στο πλαίσιο του μορατόριου, εντό εισαγωγικών έτσι, και στο Δίνεκε να παρέμειναν κλειστά 8, που υποθέτω ότι αυτό είναι εφικτό, αυτό σημαίνει ότι 7 με 8% από το ενεργειακό μείγμα της Γερμανίας και 2% από την Ευρώπη ε, λείπει. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα ανεφοδιασμού. Το αποφασιστικό ερώτημα είναι, έχουμε συγκρίσιμες καταστάσεις και εξελίξεις σε άλλα κράτη. Αυτό το παρακολουθούμε. Ακόμα και αν οι εξελίξεις αυτές θέλουμε να συμπεριληφθούν ε, στον ενεργειακό μας οδικό χάρτη σε διάφορα σενάρια και εναλλακτικές προτάσεις για το διάστημα 2020 και επέκεινα δεκαετίες. Και στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας ε, παρακολουθούμε αυτή τη συζήτηση με πολύ προσοχή και εγώ θεωρώ ότι πουθενά σε κανένα άλλος, ε, άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα υπόλοιπα 14 που έχουν πυρηνική ενέργεια δεν γίνεται συζήτηση όπως στη Γερμανία για ε, πιο γρήγορο κλείσιμο και περιορισμό στο χρόνο λειτουργίας των εργοστασίων. Στη Γαλλία, επί παραδείγματι, δεν βλέπουμε καμία διαφορά, καμία αλλαγή, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ισπανία, για παράδειγμα, όπου ε, είναι ουσιαστική και ε, άξια αναφορά στη συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Στην Ελβετία βλέπουμε αλλαγή Στην Ιταλία έχει σταματήσει ο καθορισμός το που θα είναι εργοστάσια για ένα-δύο χρόνια. Στην Πολωνία όμως για παράδειγμα ο σχεδιασμός για ένα πυρηνικό εργοστάσιο συνεχίζει ε, χωρίς αλλαγή. Δηλαδή τώρα ανεξάρτητα από το θέμα τι θα μπορούσε κανείς να επιθυμεί επί και τι προτιμάει. Προς το παρόν δεν βλέπουμε έτσι, ουσιαστικές αλλαγές τις ποσότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ρωτήσατε ε, για το κόστος, το πλήρες κόστος και πώς υπολογίζεται αυτό. Στην πυρηνική ενέργεια στην αρχή, πριν από 50 και 40 χρόνια, η έρευνα ήταν σε μεγάλο βαθμό δημόσια και με δημόσια χρηματοδότηση και επιχορήγηση. Και το θέμα της ευθύνη αυτό τον καιρό είναι έτσι ρυθμισμένο ώστε στην χείριστη περίπτωση, ας πούμε όταν έχουμε μεγάλη καταστροφή, ε, υπάρχουν υποχρεώσεις ασφάλισης και στα κράτη-μέλη. Τα έχουμε αναλύσει αυτά έτσι σε συντομία και η μεγαλύτερη ευθύνη ε, είναι στη Γερμανία 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ευθύνη έχουν όλες οι εταιρείες ε, με το κεφάλαιό τους και τα περισσοκά του στοιχεία, αλλά και το κεφάλαιό τους ε, στο χρηματιστήριο. Ε, σε περίπτωση έτσι, χειρότερης, του χειρότερου σενάριου είναι αρκετά περιορισμένο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πυρηνικά απόβλητα και την τελική τους ε, αποθήκευση και πάλι χρειάζονται ε, προτάσεις και ρυθμίσεις. Αντίστροφο όμως δεν υπάρχει σχεδόν καμία μορφή ενέργειας όπου τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες να ε, χρηματοδοτήθηκε με τρόπο αξιο... αξιόλογο ο άνθρακας. Στη Γερμανία ή στην Ισπανία ας πούμε δεν θα μπορούσε να ε, γίνει εκμετάλλευσή του χωρίς κρατική ενίσχυση, η οποία όμως λύγει αυτή τη δεκαετία. Και εκτός από τους νόμους, ε, χρειάζεται πραγματικά στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενίσχυση αποτελεσματική, έτσι ώστε μετά ε, την εισαγωγή τους στην αγορά, κάποια στιγμή από μια χρονική στιγμή και μετά να μπορούν να στέκονται στα πόδια τους στον ανταγωνισμό χωρίς ε, χρηματοδότηση. Αυτό ισχύει ε, ε, για την υδροηλεκτρική ενέργεια και κάποια στιγμή για την αιωλική αλλά και για την ηλιακή όταν θα έχουμε μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή και όταν θα έχουμε πια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική. Με ρωτήσατε ε, για τον πυρηνικό φόρο, ε, nuclear tax. Κοιτάξτε, κάποιος συνάδελφός μας, πούμε, προτείνει ένα νέο φόρο ενεργειακό. Κάποιο άλλος συνάδελφος θέλει αυτές τις μέρες να μιλήσει ε, για ένα τέλος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή φορολόγηση στα αεροπορικά ειστήρια ή στην κυροζήνη. Αλλά στη ζωή μου εγώ έχω προσγειωθεί εδώ και καιρό. Για κάθε μορφή ευρωπαϊκού φόρου χρειάζεται ομοφωνία. Και είναι πιθανό ότι με 27 κυβερνήσεις για το φόρο χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών θα αντιδράσει το Λονδίνο ή κάποια στιγμή το Βερολίνο για έναν άλλο φόρο. Κάποια κυβέρνηση θα βρείτε μέσα στις 27, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ε, ε, δυνατότητα επιβολής ε, φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε περιορισμένη η εφεύρεση νέων φόρων. Γι' αυτό ένας οποιοδήποτε ενεργειακός φόρος, ανεξάρτητα με τη μορφή της ενέργειας, νομίζω δεν έχει ε, μεγάλες πιθανότητες, γιατί είμαστε ρεαλιστές. Για την, ε, αποθήκευση, τη δέσμευση και την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα, το CCS, μέχρι το καλοκαίρι ελπίζουμε τα κράτη να έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία και έχω ήδη ανακοινώσει στη Γερμανία. Το συζητάνε δύο χρόνια ε, το Bundestag στη Γερμανική Βουλή. του, είπα όμω ότι αν δεν δρομολογηθεί θα λάβουμε τα μέτρα μας. Και προ τα άλλα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα έξι μεγάλα μοντέλα ε, που είναι στη δική μου αρμοδιότητα, με το ένα δισεκατομμύριο που μας δώσατε για δημόσια χρηματοδότηση, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τέσσερις ε, τέσσερα ή πέντε μεγάλα σχέδια επίδειξης έχουν ξεκινήσει και πρέπει να σας πω ότι μέχρι το 2015 θα έχουμε ε, αποτελέσματα από αυτά τα μοντέλα και ε, για σας, για τη μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ήταν σημαντικά. Αρκετά σημαντικά για να έχουμε και μια μακροπρόθεσμη χρήση του άνθρακα αλλά και να αποφεύγουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε, στα βιομηχανικά κράτη και να βγάλουμε και τα απαραίτητα συμπεράσματα ε, τεχνικά, οικονομικά και πολιτικά. Το θέμα της ε, εξωτερικής πολιτικής τώρα στην ενέργεια. Πολύ συγκεκριμένα ε, συνομιλούμε με τους Ρώσους εταίρους μας και τους Ουκρανούς για να πετύχουμε ε, να υιοθετήσουν και εκείνη τις δοκιμές αντοχής. Την άλλη εβδομάδα θα έρθουν εδώ οι Ελβετοί να συζητήσουμε και ε, επίσης ε, γραπτός ε, επικοινωνούμε αυτές τις ημέρες με τις άλλες δύο χώρες που ανέφερα. Αναφερθήκατε επίσης στο λεπτό και στο θέμα της Εσωνίας, ε, Λετωνία, Λιθουανίας, Πολωνίας, Καλίνιγκρατ, Λευκορωσία, Ρωσίας. Είναι ευαίσθητο. Γιατί εσείς θέλετε και οι χώρε αυτές θέλουν να μειώσουν την εξάρτησή τους και σε φυσικό αέριο και ε, σε πετρέλαιο από τη Ρωσία. Και παίζει ιδιαίτερο ρόλο το θέμα ενός πυρηνικού εργοστασίου που σχεδιάζεται με ΑΙ ε, στη Λιθουανία. Αντίστροφο όμω και οι Ρώσοι σχεδιάζουν πυρηνικό εργοστάσιο στο Καλίνιγκραντ. Και τώρα τι γίνεται, οι Ρώσοι και οι Ευρωπαίοι θέλουμε να έχουμε ε, ανοιχτή τι δυνατότητα εμπορίου, ή ε, ε, ε, δυνατόν στον ΠΟΕ, ελευθερία, ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και προϊόντων. Για τον άφρακα το έχουμε, γιατί χρειαζόμαστε το άφρακα και, και τον εισάγουμε από τη Ρωσία. Τα ίδια για το πετρέλαιο, για το φυσικό αέριο ακόμα περισσότερο. ρεύμα ηλεκτρικό δεν εισάγουμε. Μόνο έτσι έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση που χτιστεί ένα τέτοιο εργοστάσιο στο Καλίνεγκρατ. Μπορούμε να το ζητήσουμε. Από την άλλη όμω, αν απαιτήσουμε και πετύχουμε υψηλότερη προδιαγραφή ασφαλείας στο Καλίνιγρα, τότε θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι, ας πούμε ότι θα γίνει αυτό, ξαφνικά η εξολόγηση της αγοράς για ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Λιθουανία θα ήταν τελείω διαφορετική. Είναι πόκερ όλη αυτή η ιστορία. Εγώ είμαι σε στενή ε, συνεργασία και επαφή με την κυβέρνησή σα, αλλά θα πρέπει να αποφασίσουμε είτε θέλουμε τα υψηλότερα στάνταρ να τα επιβάλλουμε στο Καλίνιγκρατ και θα ανοίξουμε την περιοχή ε, την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, είτε θα την έχουμε κλειστή και δεν θα εισάγουμε ρεύμα από τη Ρωσία, μόνο άνθρακα, αέριο και πετρέλαιο ε, και θα είναι πιο επισφαλής η κατάσταση των πυρηνικών εργοστασίων εκεί στην περιοχή και οι Πολωνοί ως άμεσος γείτονας δεν είναι τόσο σίγουροι τι θέλουν. Αν θέλουν να εισάγουν ηλεκτρικό ρεύμα από τις γειτονικές τους χώρες. Για τις δοκιμές ε, ε, αντοχής. Δεν Εμείς επιτύχαμε να το, να το αποφασίσει αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στην αρχή δεν ήταν καθόλου προφανές αυτό, ήταν πολύ μεγάλες οι αντιστάσεις και πολλές. Τώρα όλα τα κράτη-μέλη δήλωσαν προθυμία εθελοντικά να δεχτούν ε, τις δοκιμές ε, αντοχής. Και εγώ επικαλούμε τώρα και την τέχνη του εφικτού και του πρακτικού. Να είναι διαφανής η διαδικασία που θα ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη, αλλά στην ουσία εδώ περί τίνος πρόκειται. Στη συνθήκη της Λισαβόνας ορίζεται ότι το ενεργειακό μείγμα είναι ε, υπόθεση των κρατών μελών. Και το λέω έτσι με κάθε φιλικότητα. Εγώ ως μοχλός δεν έχω μεγάλη επιρροή κατά των ε, πλειοψηφιών στα εθνικά κοινοβούλια. Ό,τι δεν πετυχαίνετε εσείς στο Παρίσι, δύσκολα μπορείτε να το πετύχετε μέσω αιμού στις Βρυξέλλες. Απλώς δέχομαι, επειδή σέβομαι τους νόμους, ότι το ενεργειακό μείγμα παραμένει ε, υπόθεση των κρατών μελών, δεν έχει αλλάξει. Παρά αυτό δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη με το θέμα αυτό, γιατί καταφέραμε τη μεγάλη καμπή, το 20% ανανεώσιμες ενέργειες, σε 9 χρόνια. Είμαστε υποχρεωμένοι. Με εκθέσει προόδου επίσης το ελέγχουμε, είμαστε σε καλό δρόμο. 20% σημαίνει ότι μόνο 80% μετά από το ενεργειακό μείγμα είναι υπόθεση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ας αφήσουμε στην άκρη το πετρέλαιο και τις μεταφορές. Και πάμε σε αυτό που μας ηλεκτρίζει όλους, που είναι η ηλεκτρική ενέργεια. 20% ανανεώσιμες σημαίνει και 35% αιωλική ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια, η υδροηλεκτρική, η βιομάζα ή δεν ξέρω τι άλλο. Ε, δηλαδή, σε νέα χρόνια θα έχουμε 35% του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται στα κράτη-μέλη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε, για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τα επόμενα τρία χρόνια θα έχουν ξεπεράσει ανανεώσιμες τον άνθρακα και σε 4-5 χρόνια και την πυρηνική ενέργεια. Και από το 2016 θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό και με τον οδικό χάρτη ε, τολμούμε και μία πρόταση, γιατί η ασφάλεια του σχεδιασμού και του προγραμματισμού είναι απαραίτητη στην ενέργεια. Οπότε ε, με τα βεβαιότητα στο 2025 και το 2030 θα φτάσουμε στο 40% και παραπάνω στην ηλεκτρική, επαναλαμβάνω, ενέργεια θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Και με κάθε ποσοστό που συμφωνούμε δεσμευτικά στην Ευρώπη, μειώνεται το ποσοστό που έχουν στην ίδια τους, ε, τη διακριτική ευχαίρεια τα κράτη-μέλη. Ακόμα περισσότερο. Δηλαδή είναι μια διαδικασία ε, το άρθρο 194 ε, όλο και περισσότερο εκχωρείται και η απόφαση και ο έλεγχος στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτή η μεγαλύτερη καμπή ε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό θα γίνει όταν θα πετύχει το πακέτο μας για τις υποδομές. Ένα πανευρωπαϊκό πακέτο στην ηλεκτρική ενέργεια και με δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας. Θα θυμάστε ότι εσείς ήδη πριν από ένα εξάμεινο ψηφίσατε την οδηγία για ε, τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Θα πρέπει να έχουμε αποθηκευμένο για 30 ημέρες φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Εγώ μηχανικός δεν είμαι, αλλά κάπου έχω ένα όραμα στην ίδια μας τη γενιά να έχουμε μια οδηγία και για το ηλεκτρικό ρεύμα και τον εφοδιασμό. Και να έχουμε ας πούμε 30 μέρες ε, αποθηκευμένο το ρεύμα σε διάφορες μορφές, ε, ε, ε, μορφή μεθανίου, υδρογόνου, συμπιεσμένου αερίου, βιολογική ενέργεια, ό,τι θέλετε. Και εμένα είναι όριμο αυτό. Να προχωρήσει τόσο πολύ η έρευνά μας στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και να μπορούμε σε ένα ορατό μέλλον να έχουμε αυτή την ανεξαρτησία των 30 ημερών όπως έχουμε για το φυσικό αέριο ή ακόμα και για το πετρέλαιο που είναι 110 ημέρες η ε, αυτονομία μας, ας πούμε, με την αποθήκευση. Και στον άνθρακα το έχουμε και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο, ας το έχουμε και στον ηλεκτρισμό. Ευχαριστώ πολύ κύριε πίτροπε. Είκοσι λεπτά χρειαστήκατε για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Είμαστε λοιπόν στις 5 παρα 2 λεπτά. Και τέλειωσε ο χρόνος μας. Λυπούμε βεβαίως για όλες και όλους εκείνους τους συναδέλφους που δεν πρόλαβαν να θέσουν ερωτήσεις. Πάντως νομίζω άξιζε τον κόπο η συζήτηση αυτή. Ακούσαμε πολλά και σημαντικά πράγματα. Το θέμα θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Η Επιτροπή μας θα συζητήσει ιδιαίτερα τον οδικό χάρτη ενέργειας του, μέχρι το 2050 διότι ακριβώς αυτά που είπατε για τις ανανεώσιμες ενέργειες, τις οποίες πάντοτε εμείς έχουμε υποστηρίξει όσο περισσότερες τόσο καλύτερα και γι' αυτό και ένα ενεργειακό μέλλον το οποίο σίγουρα θα είναι πιο καθαρό και ελπίζω παρόλα αυτά να διατηρείται σε σχετικά χαμηλό κόστος. Οι εξαγωγές πετρελαίου μιλήσατε για τις προθεσμίες και βέβαια για την αποδοτική ενέργεια, την αποδοτικότητα μάλλον της ενέργειας, είπατε επίσης τα σχετικά, καθώς επίσης και τις ε, προθεσμίες για την βολή προτάσεων. Τώρα, θα επανέλθουμε όπως είπατε σε διάλογο πριν από τα μέσα Μαΐου για τα κριτήρια των δοκιμασιών αντοχής. Σας ευχαριστώ πολύ και θα σας ξαναειδώμε. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann äh, Βρισκόμαστε λοιπόν μέσα στα όρια του χρόνου μας. Διότι δυστυχώς νόμιζα ότι θα μπορέσει να υπάρξει και δεύτερη, ε, δεύτερος γύρος. Ορισμένοι συνάδελφοι όπως η Λίντα Μακάβαν, ο Καλ Χάιντς Φλόρεντς είχαν ακόμη ζητήσει το λόγο. Δεν ήθελα να διακόψω τον Επίτροπο στις απαντήσεις του. Δυστυχώς ο χρόνος πέρασε. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα τώρα που είναι η έκθεση της Dagmar roth για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μεταδιδόμενες πογκώδεις εγκεφαλοπάθειες και τους σχετικούς ελέγχους ζωοτροφών και τροφίμων. Θα μας εξηγήσει με λεπτομέρειες βεβαίως η Dagmar Roth-Berend. Έχετε το λόγο Dagmar. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μεταδιδόμενες πογκώδεις εγκεφαλοπάθειες. Τέλος πάντων, ενσεφαλόπαθη, ας το πω έτσι, ε, λέγεται στα αγγλικά και είναι εγκεφαλοπάθεια. Τέλος πάντων, ε, λίγο έχω μπερδευτεί, το έχω πει τόσες πολλές φορές την λέξη αυτή τα τελευταία 15 χρόνια. Μιλούμε λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μια έκθεση για το δεύτερο οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όχι μόνο τις ε, σπογκώδεις εγκεφαλοπάθειες των βοηδών. Κουν Φαντάχ είσαι κάπου εδώ της Επιτροπής. Θα μπορούσε να με βοηθήσει με την προφορά αυτής ε, της ορολογίας. Τέλος πάντων μιλούμε για όλο το φάσμα, δηλαδή και ε, άλλων ζώων όπως εγών, προβάτων, ιδίως, ιδίως. Θεωρητικά μπορούν να πλήγονται, να πλήττονται συγγνώμη, και άλλα ζώα από τις νόσους αυτές. Πάντως, από την νομοθεσία μας του 96-97-98 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φτιάξει ήδη ένα roadmap το 2005 όπου έκανε μια προσπάθεια να εγκύψει στην τότε κατάσταση και να προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις. Τώρα έχει υποβάλει νέο roadmap η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έκθεση αυτόν τον roadmap έχει ως αντικείμενο. Πρώτα, οι οδικοί αυτοί χάρτες έχουν τον στόχο πάντοτε αφενός να εγκύψουν στο ερώτημα πώς διεξάγονται τα τεστ του BSE, το, ποια θα πρέπει να είναι η ηλικία των ελεγχόμενων ζώων, ποια είναι τα, ε, το, το ενδεχόμενο επικίνδυνο υλικό, πώς αφαιρείται αυτό και ούτω καθεξής. Αυτά πάλι είναι τα κεντρικά θέματα της, ε, του νέου οδικού χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ μάλιστα προστίθεται και το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της αναφέρεται και στην ισχύουσα απαγόρευση ε, χορήγησης στα ζώα ε, ζωικών αλεύρων από μη μυρικαστικά σε, μη, σε μυρικαστικά. Υπάρχει για την ώρα πάντως ξεκάθαρη νομοθεσία παράτημα 5 της ε, σχετικής οδηγίας. Υπάρχει λοιπόν η σχετική νομοθεσία για τα θέματα αυτά, την οποία τηρεί απολύτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την σύνταξη του καταλόγου των επικίνδυνων υλικών θα υπάρχει μάλλον και σημείωμα η ανακοίνωση της ΕΦΣΑ θα υπάρξει μάλλον γιατί για την ώρα η ΕΦΣΑ δεν αλλάζει την θέση της όπως και εγώ άλλωστε το απλούστερο βέβαια είναι να έρθω στην ίδια την έκθεση και στα ιδιαίτερα θέματα του οδικού χάρτη πρώτα πώς κρίνω συνολικά τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι όπως μέχρι τώρα πραγματικά είναι καλό το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως δεν συμφωνώ πάντοτε και σε όλα, κάτι τέτοιο θα ήταν και περίεργο, αλλά αντίθετα από παλαιότερα, αντίθετα με παλαιότερες Ευρωπαϊκές Επιτροπές της δεκαετίας του 90, όπου τίναμε μάλλον να φοβούμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργαζόταν ε, πίσω από την πλάτη μας με τις χώρες μέλη. Στην παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πράγματα έχουν αλλάξει και γι' αυτό ο δικός χάρτης που υποβάλλει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της BSE είναι εντάξει. Βεβαίως θα εξετάσουμε και τα επιμέρους θέματα. Υπενθυμίζω ότι μιλούμε για μεταδοτικές σπογκώδεις εγκεφαλοπάθειες, κυρίως βοηθών αλλά και εγώ προβάτων, λιγότερο βεβαίως. Μιλούμε για το 2009 για παράδειγμα όπου έγινε μια καταγραφή για 69 περιπτώσεις συνολικά. Πρώτα πρώτα λοιπόν η παρατήρηση των, των, ε, της πορείας της εγκεφαλοπάθειας. Αυτά είναι οι παράγραφοι 3, 3, 3 έως 6. και πρόκειται για εξέταση βοηδών άνω των 72 μηνών ηλικίας από ε, διάφορες χώρες μέλη. Στην διαδικασία της επιτροπολογίας την έχουμε εξετάσει. Συζητήσαμε αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Εγώ τότε όταν το συζητήσαμε αυτό είχα την αίσθηση ότι μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε την αύξηση του ορίου ηλικίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το ετήσιο πρόγραμμα παρακολούθησης της BSE έχει εκπονηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε γίνεται μια προσπάθεια σωστής καταγραφής των διαφόρων ελέγχων. Το δε πρόγραμμα παρακολούθησης της BSE επικαιροποιείται τώρα με την αύξηση του ορίου ηλικίας. Είπα και πάλι ότι έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφερθεί και στις όπως είπα πριν, είναι ορισμένες χώρες μέλη, δηλαδή 22 συνολικά. Οι 5 λείπουν, οι 5 αυτές χώρες μέλη λείπουν, δηλαδή Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Λείπουν από την καταγραφή αυτή. Μπορούμε να τα περιλάβουμε εφόσον γίνει η αύξηση του ηλικίας και στις υπόλοιπες 22 χώρες, εάν υπάρχει μια συνολική καταγραφή των κινδύνων, κάτι το οποίο δεν γίνεται, δεν υπάρχει ακόμη. Ο λόγος είναι ότι σε ορισμένες από τις νέες εντός εισαγωγικών χώρες μέλη μπόρεσε να εξασφαλιστεί πολύ ιστερότερα η εφαρμογή της απαγόρευσης χορήγησης ζωοτροφών ζωικής προέλευσης σε μη μυρικαστικά. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να εξακολουθήσει να γίνεται μια διάκριση. Αυτή η διάκριση γίνεται καταφανής εν προκειμένως και στη διαφορετικές ηλικίε των εξεταζόμενων ζώων. Έχει καλώς. Και ούτε το αμφισβητούν οι ενδιαφερόμενες χώρες. Δυσκολεύομαι πάντα λίγο να δεχθώ ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ριου ηλικία στον έλεγχο των βοηδών, διότι εξακολουθούν και υπάρχουν περιπτώσεις, αν και βέβαια σε χαμηλότερη ηλικία σχεδόν ποτέ, το 2009 δηλαδή έχουμε μία μοναδική περίπτωση στην Τσεχία στην ηλικία 48-59 μηνών μεταξύ των πέντε προαναφερθιστών χωρών. Οι περισσότερες κατά τα άλλα περιπτώσεις BSE είναι σε ζώα που εσφάγησαν γη ή σε ζώα τα οποία ε, βρήκαν τον θάνατο με διαφορετικό τρόπο και άνω των 60 μηνών. Αυτό είναι αυτονόητο και εξηγείται και από το ιστορικό. Όσο πάντως εξακολουθούμε και έχουμε περιπτώσεις BSE, νομίζω ότι πρέπει να διατηρούμε, να τηρούμε μάλλον τα όρια αυτά ηλικία και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και για τις ε, έρευνες θα γίνονται από τον Ιανουάριο του 2013 και μετά. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε ιδιαίτερα είναι βέβαια η παράγραφη 7 έως 13 της εκθεσής μου που αναφέρονται στην παραπέρα απαγόρευση χορήγησης ζωοτροφών ζωικής προέλευσης. Πριν από πολλά χρόνια αποφασίσαμε να επιβληθεί απαγόρευση χορήγησης λευκόματος ζωικής προέλευσης σε μη μερικαστικά, δηλαδή χοιρινά, πουλερικά. Χοιρινά και πουλερικά στην αγροτική εκμετάλλευση είναι πανφάγα ζώα. Τα τρώνε, τρώνε τα πάντα και τους χορηγούνται τα πάντα. Είναι και τα ζώα τα οποία παλαιότερα λάμβαναν ως ζωοτροφή ζωικά άλευρα. Ζωικά άλευρα, δηλαδή από κατάλοιπα ζώων, σφαγίων, που ήταν υποτίθεται κατάλληλα για, ανθρώπινη, για από ανθρώπους. Όχι ωστόσο ολόκληρο το ζώο. Δηλαδή εμείς τρώμε ίσως το μισό του ζώου περίπου από, από ένα ζώο περίπου το 50%. Σε, ο, ορισμένα στα βοηθή είναι λίγο περισσότερο, στα χοιρινά είναι λιγότερο. Και το υπόλοιπο του σφαγίου γινόταν παλαιότερα ζωικό άλευρο. Από την εποχή της πουγκόδους εγκεφαλοπάθειας, ωστόσο και μετά, που προέκυψε από το γεγονός ότι δόθηκε σε μυρικαστικά μολυσμένο ζωικό άλευρο, μυρικαστικά τα οποία είναι φυτοφάγα ζώα. Έτσι λοιπόν υπήρξε αυτή η, θα έλεγα, συναισθηματική απέτηση του κοινού, γιατί βέβαια επιστημονική, θε, επιστημονική θεμελίωση δεν υπάρχει, ούτως ή άλλως η χορήγηση ζωικών αλεύρων σε ε, μυρικαστικά απαγορευόταν ούτως ή άλλως. Και αυτό το πρόβλημα που προέκυψε ήταν διότι δεν ήταν επισημασμένα τα ζωικά αυτά άλευρα. Βέβαια στην αγροτική εκμετάλλευση ανα πάσα στιγμή εξακολουθεί να είναι δυνατόν να χορηγηθούν τέτοια ζωικά άλευρα και σε βόηδη. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει να προκαλείται πρόβλημα. Και οι αγρότες ούτως ή άλλως έχουν παραδοσιακές αντιλήψεις σε ό,τι αφορά την ε, προστασία και ευημερία των ζώων τους. Ψάχνω να βρω με το βλέμμα την κυρία Πάουλσεν, την οποία είδα προηγουμένως, και ο κύριος Νέλχαρτ έχει κάνει πολλά για, την, ε, για τον ελέγχο της υγιεινής και την επικινδυνότητα ορισμένων συστημάτων κλπ. Για πολύ καιρό λοιπόν μπορέσαμε να αποφύγουμε την χρήση σημαντικών ποσών ε, ζωικού λευκόματος ε, που απευθυνόταν σε ζώα τα οποία μπορούν να φάνε κάτι τέτοιο. Θυμάστε και την έκθεση Χόισλινγκ για την έλλειψη ζωικού λευκόματος και με γνωμοδότηση για τη δική μας επιτροπή του κ. Ταμπάτσι. Και το συμπέρασμα ήταν ότι δεν διαθέτουμε επαρκές ζωικό λεύκομα για, με προσμού ζώα τα οποία το χρειάζονται και ιδιαίτερα τα ζώα που ανέφερα πριν που είναι παμφάγα. Το ίδιο συμπέρασμα ήταν επίσης ότι η εναλλακτική επιλογή, δηλαδή να δίνεται γενικά τροποποιημένη σόγια, ήταν δυσχερής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα προτείνει βέβαια πολύ προσεκτικά και επιφυλακτικά μια επανεξέταση της απαγόρευσης χορήγησης τέτοιων ζωικών αλεύρων και το προτείνει με κάποια επιφύλαξη διότι γνωρίζει πόσο συναισθηματικά φορτισμένο είναι το θέμα. Το γνωρίζω και εγώ βεβαίω. Και παρόλα αυτά είπα ανέκαθεν ότι ωραία είναι τα συναισθήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δικαιολογημένα, αλλά εδώ εμείς έχουμε πολιτική εργασία να κάνουμε και νομοθετική εργασία και δεν θα πρέπει να παρασυρώμεθα μονάχα από συναισθήματα. Γι' αυτό προτείνω υπό ορισμένε προϋποθέσεις να επιτρέπεται η χορήγηση ζωικών αλεύρων στα ζώα που μπορούν να το καταναλώσουν και αυτό βεβαίως υπό ορισμένε προϋποθέσεις. Βλέπω ότι ο κύριος Σνέλχαρτ έχει ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για τα όσα είπαμε τα σχετικά με το συνέστημα και τη συναισθηματική φόρτιση. Απάντηση χωρίς μικρόφωνο από άλλη Ευρωβουλευτή. Καλώς λοιπόν, ευχαριστώ. Το προτείνω, όπως είπα, οι ορισμένε προϋποθέσεις, υπό όρους. Αφενός προτείνω να διασφαλίζεται η εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών για την παραγωγή των ζωικών αλεύρων. Προ 13 ετών νομίζω, δηλαδή το 1998-99, εκεί περίπου είχαμε εγκρίνει νομοθεσία για παραγωγή με μέθοδο υψηλής πιέσεως και θερμοκρασίας, που εξακολουθεί και είναι η, η βασική απέτηση το gold standard ας πούμε στην βιομηχανία. Βλέπω βεβαίω και τους προσώπους της Κομισιόν εκεί που νεύουν καταφατικά. Αυτή η μέθοδος προβλέπει ότι τα υπόλοιπα των ζών προβλέπεται να περάσουν για ένα ορισμένο διάστημα, 10 λεπτά νομίζω, με κάποια πίεση ε, υψηλών πολλών μπαρ και υψηλή θερμοκρασία. Αυτό όταν ακόμα επιτρεπόταν η χορήγηση τέτοιων ζωικών αλεύρων. Υπήρχε η δυνατότητα τότε βεβαίως με λήψη τμήματων μόνο υγιών σφαγίων, των οποίων το κρέας κατευθυνόταν στην κατανάλωση, να ε, παραχθεί ζωικό αλεύρό. Λοιπόν, εγώ προτείνω τη χρήση αυτής της μεθόδου. Επίσης προτείνω απαγόρευση του κανιβαλισμού, δηλαδή διατήρηση της απαγόρευσης του κανιβαλισμού. Και εδώ βεβαίως πρόκειται για θέμα λίγο πολύ συναισθηματικής φόρτισης. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να υπάρξει και cross-contamination, αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό όταν ε, χείρι καταναλώνουν χείριο κρέας. Παρ' όλα αυτά, ας, εξακολουθήσουμε, ας εξακολουθήσει να ισχύει η απαγόρευση ώστε να, να αποφευθεί και η τελευταία, το τελευταίο ενδεχόμενο της λεγόμενης cross-contamination. Εξαιρούμε ρητά τα βοηθή. Γιατί, ρώτησα, ή με ρώτησαν. Και η απάντηση ήταν, διότι αυτό προσφέρει ακόμα μια εγγύηση, ακόμα υψηλότερη εξασφάλιση δηλαδή, εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με ορισμένα προϊόντα. Εάν εξασφαλίσουμε επίσης διαχωρισμό των οδών μεταφοράς και παραγωγής και ε, αντίστοιχη επισήμανση, τότε αυτό που προτείνω μπορεί να είναι μια, ένα άνοιγμα μιας θύρας για την επαναλήψη της χορήγησης ζωικών αλεύρων σε ζώα τα οποία μπορούν να τα καταναλώσουν. Όχι βέβαια για διατροφή κατοικιδίων. Βέβαια πρέπει να είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τον έλεγχο και των ζωικών πρωτεϊνών ώστε να είναι σαφές ότι ε, τηρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσει. Τονίζω επίσης στην έκθεσή μου ότι δεν μπορεί να υπάρξει εισαγωγή ορίου ανοχής για τη χορήγηση ζωικών αλεύρων σε μυρικαστικά ζώα. Τώρα οι παράγραφοι 13 και 14 της εκθεσή μου εγώ λέω ότι αναμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην λίστα να περιλάβει και να μην οδηγήσει σε οποιαδήποτε αποδυνάμωση από πλευράς του Διεθνούς Γραφείου Επιζωτιών. Υποστηρίζουμε και ορισμένε έρευνες τώρα για την ανθεκτικότητα στα εγωπρόβατα. Εγώ είπα ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εξάλληψη των περιπτώσεων ε, εγκεφαλοπάθειας. Ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει ό,τι αφορά την εξέταση επιζών των ζώων. Έχω ε, θέσει τώρα και ορισμένα θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη 19-22 παραγραφή μου όπου τονίζω ότι υπάρχει, διαμορφώνεται μια θετική τάση για την αναγνώριση περιπτώσεων BSE και για την δημιουργία ενός συστήματος εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενό συστήματος ε, ε, δοκιμασιών ότι το σύστημα που υπάρχει είναι σωστό αλλά σε ορισμένες χώρες μέλη εξακολουθεί η ποιότητα να είναι χαμηλή και αυτό λέει στην παράγραφο 2 της έκθεσης της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους επίσημους ελέγχους ορισμένων κρατών μελών. Ένα από τα πιο αγαπητά μου θέματα που το έθιξα ήδη είναι στις παραγράφους 23-25. Πρόκειται για κρέας το οποίο έχει ανακτηθεί με μηχανικό τρόπο, δηλαδή έχει διαχωριστεί από τα οστά. Εγώ θα ήθελα να παραμείνει απαγόρευση, γιατί έχουμε αρκετό κρέας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται να αποχωριστεί και η τελευταία ίνα ε, σάρκας από τα οστά. Τέλο πάντων αυτό μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον για ορισμένα είδη αλλαντικών. Και εν τέλει είμαι πεπισμένη ότι οι νομικές διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή στις χώρες μέλη για το κρέας αυτό έχουν καλώς και ο στόχος θα πρέπει να είναι να εξεταστούν οι ορισμοί και εγώ επιθυμώ να εισαχθεί και επισήμανση διότι πιστεύω ότι πολλοί καταναλωτές δεν θα αγόραζαν. Τώρα για, τους, για τις διοξίνες στα ηχθιάλευρα. Οι τιμές ε, κατοφλίου είναι, ε, μάλλον οι ανώτατες τιμές είναι πολύ υψηλές και κυρίως υπακούν σε σκοπιμότητες και όχι σε μια πραγματική ε, προστασία της ανθρώπινης υγείας και της υγείας των ζώων. Κυρίως τίνουν στην διασφάλιση κάποιων αλλιών από την ε, Βόρεια Θάλασσα. εκεί πρέπει να διατηρηθούν και οι διατάξει υγειονομική προστασία. Αυτό τα έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Σνέλχαρτ που έχει κάνει και τι σχετικέ εκθέσει παλαιότερα. Και εφόσον ε, χρησιμοποιούνται τέτοια ζωικά άλευρα πρέπει να είναι αποστηρωμένα. Και τέλος η παράγραφος 18, η καταστροφή ομάδων ζώων, εφόσον σε μια αγέλη εμφανιζόταν μία περίπτωση σπογκώδους εγκεφαλοπάθειας τότε θα ανατώνεται ολόκληρη η ομάδα και μόνο εφόσον η ενδιαφερόμενη χώρα μέλος ζητήσει να διατηρηθεί στη ζωή η συγκεκριμένη ομάδα μέχρι τέλους της παραγωγικής ζωής της αλλά να μην χρησιμοποιηθεί το, κρέα, το κρέας της για παραγωγή κρέατος, τότε αυτό ενδεχομένω να γίνεται δεκτό. Τώρα κάνει μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία όμως εγώ απορρίπτω απολύτω και είναι και το μοναδικό σημείο το οποίο απορρίπτω, αλλά για τους αρμοδίους κυρίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη. Εγώ θεωρώ ότι η κατάσταση όπως διαγράφεται επί του παρόντος εξακολουθεί να δικαιολογεί την ε, καταστροφή των αγελών που κινδυνεύουν από ε, κεφαλοπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, εν το συνόλο της η έκθεση είναι ε, σφιχτή, είναι σύντομη, είναι βεβαίως πλήρης ε, πληροφοριών με ε, υποστήριξαν θαυμάσια οι συνεργάτες και της, Ευρωπαϊκής... και της γραμματείας μας που δεν είχαν και γνώση προτέρα του θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία. Ευχαριστώ για την συνεργασία λοιπόν και την ε, Γραμματεία της Επιτροπής και τη συνεργάτη μου που κάθεται πίσω. Euh, euh, Ευχαριστούμε την κυρία Ροντ Μπέρεντ για αυτήν την πολύ ισόρροπη έκθεση. Θα δώσω τώρα το λόγο στους ε, εισηγητές, ξεκινώντας από τον κύριο Στάινχαρτ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να έχουμε ένα δεύτερο δρομολόγιο τώρα ε, πρόγραμμα παρακολούθησης των ε, μεταδοτικών σπογγοειδών εγκεφαλοπαθειών και όχι μόνο στα βοηθή. Τα τελευταία χρόνια μας απασχόλησαν πάρα πολύ και αν δούμε τι έχει γίνει από το 1990, όπου έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάρα πολύ γρήγορα αλλάξαμε τις διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει τώρα ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά διαπιστώνουμε πάρα πολύ ε, έντονα ότι ε, μειώθηκαν ταχύτερα τα κρούσματα και έχουμε μια τελείως διαφορετική πλέον κατάσταση και θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Τα θετικά αποτελέσματα μήπως πρέπει να βρουν και την νομοθετική ε, οδό έτσι ώστε να μην έχουμε τόσο αυστηρή ρύθμιση πλέον που έχει ξεπεραστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν χρειάζεται. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ε, την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και των ζώων και της υγείας τους. Γι' αυτό πιστεύω ότι η πρόταση της συζυγητριάς μας είναι εύστοχη ε, σε πολλούς τομείς. Για τα θέματα της παρακολούθησης για τη ΣΕΒ, τη σπογκώδη κεφαλοπάθεια των βοηθών, εγώ δεν ήμουν τόσο αυστηρός, δεν το βλέπω τόσο αυστηρά ε, για τον περιορισμό της ηλικίας. Τα τελευταία χρόνια κάναμε πολύ πολλές έρευνες και είναι και δαπανηρό αυτό. Απλώς θέλω να πω το εξή ότι το κόστος εδώ δεν είναι γνώμονας για την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν σκέφτομαι το οικονομικό κόστος εκεί, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα πολλές μελέτες και έρευνες που δεν επιφέρουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Για την αύξηση της ηλικία, εγώ θα ήμουν αρκετά γενναιόδωρος θα το ξανακοιτάξουμε. Δεν είμαι τόσο αυστηρός εγώ όσο η συγγήτρια. Πάντως θα πρέπει να συνεννοηθούμε, να δούμε τι είναι δυνατό και τι αδύνατο. Και τι είναι εφικτό και τι ανέφικτο. Ωραία. Να το ξανασυζητήσουμε αυτό το σημείο της ηλικία. Τώρα, για την απαγόρευση χορήγησης ζωοτροφών. και το θεωρώ ως κέντρο βάρους της δικής μου δουλειάς. Πρόσφατα εγκρίναμε τον κανονισμό για τη ζωική διατροφή, τη διατροφή των ζώων. Και μπορούμε να υιοθετήσουμε από εκεί κάποιες κατηγορίες, κατηγορία 3 ας πούμε των υποπροϊόντων ή των παραπροϊόντων. Και βέβαια συμφωνώ, τα σφαγεία θα πρέπει να ελέγχονται, να έχουν έγκριση και άδεια και να είναι καλή η μεταφορά και ασφαλής. Βεβαίως όλα αυτά και να αποκλείεται ο κανιβαλισμός, δηλαδή να ταΐζουμε ζώα, ε, με ζώα του ιδίου είδους ε, και στο μέλλον να φροντίσουμε τα μυρικαστικά να μην τρώνε ζωικές πρωτεΐνες. Αυτό να το σημειώσουμε και να, και να το ε, καθορίσουμε για πάντα. και ανατομικά και φυσιολογικά και ψυχολογικά δεν είναι σκόπιμο ούτε ευσταθεί κάτι τέτοιο. Και να το ορίσουμε αυτό να ισχύει και να μην το ξανασυζητήσουμε. Ωστόσο, ε, χρειάζεται και αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε ε, κατά πόσο ε, να βάλουμε μια ανοχή έστω και χαμηλή στη διατροφή των μυρικαστικών. Αυτό έχει να κάνει με τις μεθόδους παραγωγής. Δηλαδή, να μην έχουμε εσκευμένη ε, ανάμιξη ζωικών πρωτεϊών, αλλά υπάρχουν μέθοδοι παραγωγής στη βιομηχανία που ε, μοιραία δεν μπορεί να αποφευθεί η συμπέριληψη ζωικών πρωτεϊνών. Και αυτό που θέλω να το αναφέρουμε. Κάτι άλλο για την έρευνα. Συμφωνώ με την κυρία Ροτ και θα ήθελα να ακούσω με ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έγινε, γιατί πριν από χρόνια, θα θυμάστε, την πρώτη αλλαγή που είχαμε αποφασίσει εδώ για την έρευνα, για τα πρόβατα, να ε, προσπαθήσουμε με μεθόδους ε, εκτροφής, ζωοτεχνίας, ε, να μειώσουμε τον κίνδυνο. Τι έγινε με αυτό. Για τη σφαγή ολοκλήρων ομάδων ή αγελών, και εγώ δεν συμφωνώ Και δεν μπορούμε και από πλευρές προστασίας των ζώων να το ζητάμε και με το ε, ζωικό κεφάλαιο που έχουμε, ολόκληρες αγέλε να σφαγιάζονται επειδή αρρώστησε ένα ζώο. Ξέρω, δεν έχουμε πλέον οξέα περιστατικά και κρούσματα, απλώς διαπιστώνονται σε κάποιες ε, εξετάσεις. Ε, λοιπόν, να ε, χαλαρώσουμε αρκετά τα πράγματα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται η κατάσταση και να προσαρμοστούμε περισσότερο στην πραγματικότητα. Τώρα, υπάρχει και ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Τι γίνεται με τις διοξίνες και τα βιολογικά αέρια. Τι δουλειά έχουν εδώ αυτά, σε αυτό το ψήφισμα. Είμαι λίγο διχασμένος. Προσωπικά θα θεωρούσα όχι, αλλά το συζητάω. Ε, για τα διοξίνες όταν ζητούμε να αλλάξουν οι ανώτατε τιμέ. θυμάστε, το 1990, όταν ξέσπασε, το 99, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο στο Βέλγιο, κάναμε πιο αυστηρά τα όρια. Και στη ρήπανξη που ε, έχουμε από εγκαταστάσεις καύσης σε διάφορα άλλα εργοστάσια δεν μπορούμε να αλλάξουμε γιατί κινδυνεύουμε να μην μας αφήνουν να βγάζουμε στο λιβάδι τις αγελάδες μας να βοσκήσουν αν είναι υπερβολικά αυστηρές ή ωραϊκές τιμές. Για το κρέας μηχανικής ανάκτησης και εγώ ξέρετε ότι ήμουν επιφυλακτικός πάντα προσεκτικός να το συζητήσουμε αν θέλετε να το απαγορεύσουμε ας το προσπαθήσουμε και αυτό. Ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα θα το θεωρούσα υπερβολικό. Η σήμανση άλλο, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τη σήμανση. Κατά τα πιστεύω ότι είναι καλή η έκθεση που μας παρουσιάζεται, ε, περιλαμβάνει τα νέα δεδομένα και ε, ξεκονομούμε και κόστος χωρίς να απειλείται η ζωή του των ανθρώπων ούτε των ζώων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που κυρία Στελχάρτα. Πόλσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. είναι σχεδόν ιστορία πια και γι' αυτό είναι και πολύ ενδιαφέρον να διαβάζει κανείς αυτό το έγγραφο. Ήμουν μέλος της Επιτροπής αυτής και τότε ασχολούμασταν με τους ελέγχους των τροφίμων, την υγιεινή των τροφίμων επί σειρά ετών. Είχαμε αυτές τις συζητήσεις και θυμάμαι, μάλλον πάντοτε παράγει πολύ καλά κείμενα η κυρία Μπέρεντ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το κείμενο αυτό καθεαυτό. Νομίζω όμως ότι έχει έρθει η ώρα να αναγνωρίσουμε ε, ότι αντιμετωπίζουμε έλλειψη διαθέσιμων ζωοτροφών με περιεκτικότητα σε ζωική πρωτεΐνη. Αναμφίβολα η χείρη, τα, πουλερικά ε, είναι πράγματι κατηγορίες παμφάγων ζώων. Πραγματικά τρώνε τα πάντα, τρώνε ό,τι βρουν μπροστά τους. Ε, αν και βασι, κατά βάση είναι χορτοφάγα ζώα. Εντάξει, είναι όμως παμφάγα ζώα. Οπότε ε, Είμαι και εγώ υπέρ της απαγόρευσης του κανιβαλισμού. Νομίζω ότι πρέπει να, κυκλο... να απαγορευτεί η κυκλοφορία της πρωτεΐνης, της ζωικής πρωτεΐνης εντός του ίδιου ζωικού είδους. Αλλά δεν είμαι βέβαιη για το κατά πόσο έχουμε μεθόδους να διακρίνουμε μεταξύ των ζωικών πρωτεϊνών. Γιατί θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε κάποιο είδους ε, επιθεώρηση στο τέλος της αλυσίδας παραγωγής. Είναι δύσκολο να διατηρούμε διαχωρισμένες τις ζωικές πρωτεΐνες. Θα πρέπει νομίζω στο τέλος της παραγωγικής αλυσίδας των ζωοτροφών να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα ελέγχου και επιθεωρήσεων. Επίσης, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ζώων που είναι αυστηρά χορτοφάγα ε, και δεν ζουν κανένα, δεν τρώνε καμία τροφή ζωικής προέλευσης. Υπάρχει το ζήτημα της ασφάλειας των ζωοτροφών. Ε, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξει ιδιαιτέρως το ζήτημα του τρόπου πραγματοποίηση των ελέγχων στα κράτη-μέλη. Γιατί όπως είπε ο εισηγητής για τον κανονισμό, για τον, για τον έλεγχο, για τους ελέγχους, πρέπει να ομολογήσω ότι σοκαρίστηκα όταν είδα πώς γίνονται οι έλεγχοι για την ασφάλεια των τροφίμων, πώς γίνονται στην πράξη. Εμείς θεωρούσαμε ότι η αξιολόγηση του κινδύνου θα ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος ε, προσαρμογής των ελέγχων στην πραγματικότητα. Γιατί φυσικά υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών και υπάρχουν και πολύ διαφορετικά τρόφιμα που καταναλώνονται στις χώρες μέλη. Νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιτάξουμε, να ξαναεξετάσουμε το θέμα της αξιολόγησης κινδύνου. Ίσως να χρειαζόμαστε καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση, ίσως χρειάζεται να είμαστε πολύ πιο αυστηροί και πολύ πιο αναλυτικοί και εξονυχιστικοί. Ε, θα πρέπει ίσως να να ορίζουμε πολύ καλύτερα τι συνιστά κίνδυνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους επιθεωρητές να διακρίνουν μεταξύ του πολύ υψηλού βαθμού επικινδυνότητας και της σχετικής ασφάλειας. Ε, αυτά για την παράγραφο 20. Και τώρα για την παράγραφο 22. Κυρία Ροθ Μπέρεντ, ε, δεν είμαι πολύ βέβαιη πού αναφέρεστε. Ίσως θα μπορούσατε να επεξηγήσετε λίγο, να μου το επεξηγήσετε λίγο σε κατηδίαν συνάντησή μας. Ε, αυτό το μηχανικός διαχωρισθέν κρέας. Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή αν πρέπει να γελάσω. όλοι μας την καθημερινή μας ε, ζωή πετούμε πολλά φαγητά. Στη χώρα μου ο καθένας πετάει 50 κιλά εξαιρετικού κρέατος ε, στη διάρκεια του έτους. Είναι τρομερό το ποσό της, των απόλυτα φαγώσιμων τροφίμων τα οποία πετούμε. Των απόλυτα βρώσιμων τροφίμων τα οποία πετούμε. Ε, υπάρχει ανάγκη μηχανικού διαχωρισμού των, του κρέατος. Είναι ανάγκη πραγματικά να πολιτοποιούνται τα οστά ε, και να λαμβάνεται αυτό το ρευστό. Δεν καταλανώ ε, από πού πηγάζει αυτή η ανάγκη όταν τόσο πολύ φαγητό πετάγεται στο σκουπίδο τένεκε. Ποια είναι η ανάγκη να δημιουργείται αυτός ο πολιτός. όταν απόλυτα βρόσιμα τα πετιούνται. Τώρα από την άποψη της ομάδας των φιλελεύθερων αυτό που θα ήθελα να πω είναι ή μάλλον εγώ θα πρότεινα να στηρίξουμε τα μείζωνα σημεία ε, με ένα μόνο ερωτηματικό. Το ερωτηματικό μου αφορά την παράγραφο 20, το θέμα των ελέγχων και η διάρθρωση των ελέγχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ε, Nicholson. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω την έκθεση αυτή από την εισηγήτρια. Την γνωρίζω εδώ και κάποιο καιρό. Ήταν ειδικό πάνω στις κρίσεις αυτές, είτε για τη στηνόσο των τρελών αγελάδων, είτε σε άλλες κατηγορίες νόσων, επιζώτιων. Νομίζω ότι είναι το αρμόδιο άτομο για να μας κατευθύνει και νομίζω ότι η έκθεση τονίζει την σημασία της αποφυγής επανάληψης αυτού που έγινε στο παρελθόν. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα πράγματα πήγαν καλά. Αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Η σπογκώδης εγκεφαλιτήτα μπορεί να επιστρέψει, να ξαναβγεί στην επιφάνεια. Εν πάση περιπτώσει, υποστηρίζω το μεγαλύτερο μέρος ε, της έκθεσης, ε, αλλά τώρα θα ήθελα ίσως να αναφερθώ λίγο στην απαγόρευση ε, ζωοτροφών, της χρήσης ζωοτροφών σε ορισμένες, από κατηγορίες ζώων. Ε, προέρχομαι από ένα γεωργικό υπόβαθρο κατανοώ πάρα πολύ καλά τις πιέσεις, ε, το κόστος των ζωοτροφών, τι πιέσεις ασκεί στον αγροτικό κόσμο. Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε ένα μόνος τρόπος ε, να καλύψουμε το έλλειμμα της ζωικής πρωτεΐνης είναι να επιτρέψουμε αυτό το πράγμα. Ε, έχω κάποιες επιφυλάξεις. Θα επιστρέψουμε θα επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Δεν ξέρω, συμφωνώ με τα σχόλια προηγούμενων συναδέλφων επ' αυτού. Νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο που θα παρουσιαστεί το ζήτημα. Το κοινό δεν ξέρω τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, αλλά στη δική μου χώρα υπάρχει μια νοοτροπία γενική, μια άποψη η οποία αντιτίθεται στην επανεισαγωγή των ζωικών πρωτεϊνών στην παραγωγή. Συμφωνώ ολόψυχα εγώ με την άποψη της ε, εισηγήτριας, αλλά δυστυχώς θα συμφωνήσω με την κυρία Πόλσεν και θα, θα, θα πω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε το μηχανικό διαχωρισμό του κρέατος και δεν είναι ανάγκη να μόνο και μόνο για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα μερικοί άνθρωποι. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ανταποκριθούμε στο έλλειμμα των πρωτεϊνών. Ίσως αυτό φταίει η Ευρώπη, η οποία δεν αδειοδοτεί προϊόντα τέτοια από την Νότιο ή τη Βόρειο Αμερική. Ίσως αν δεν ήμασταν τόσο αυστηροί από εκεί να είχαμε λύσει το πρόβλημά μας. Φάνηκα λίγο προκλητικός σε αυτή τη δήλωση. Ομολογώ ότι αν δείτε τι γίνεται, αν δείτε τις διοξίνες, το πρόβλημα με τις διοξίνες, το οποίο συνέβη και στην δική μου εκλογική περιφέρεια. Όλα αυτά προέρχονται από άτομα τα οποία προσπαθούν να παραβιάσουν τους κανόνες και όταν τους τσακώνουν στα πράσα δεν καταλαβαίνουν γιατί ο κόσμος ξεσηκώνεται και εξαγριώνεται πρέπει όμως νομίζω να φροντίσουμε να τηρούνται οι κανόνες, πολύ αυστηροί κανόνες και προδιαγραφές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ασφαλώς μπορώ μεγάλο μέρος του περιεχομένου της έκθεσης να το στηρίξω, αλλά θα ήθελα να πορευθούμε με προσοχή και να προσέξουμε πάρα πολύ πώς θα το παρουσιάσουμε στους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Τάκμα. Ευχαριστώ. Πριν λάβουν τον λόγο οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα από τα σχόλια των συναδέλφων και πρώτα για τα όσα είπε ο κ. Σνέλχαρτ. Η αύξηση του ορίου ηλικία σε 72 μήνες ηλικία σε 22 χώρες μέλη, αυτό δεν χρειάζεται να μας απασχολήσει διότι έχει ήδη γίνει. Εγώ επισημαίνω στην έκθεσή μου ότι αυτό έχει καλώς, το έχουμε πει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ίσως υπερβολικά λογική και υπερβολικά καθώς πρέπει για να το κάνει χωρίς να ρωτήσει το Κοινοβούλιο. Αλλά αυτό που οφείλω να επισημάνω είναι ότι περαιτέρω αυξήσεις του ορίου ηλικία πρέπει να γίνουν εφόσον γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή και ότι το πρόγραμμα επιτήρησης της ε, ε, σπογκώδης εγκεφαλοπάθειας εξακολουθεί να είναι σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επί της ουσίας αλλά και συναισθηματικά όπως είπε και ο φίλος Jim Nicholson που ε, υπάρχει μια συναισθηματική φόρτιση το επιβεβαίωσε και ο ίδιος και σε αυτό εντάσσεται και ανάγκη διατήρησης της επιτήρησης της ε, BSE και εδώ εντάσσεται και το ετήσιο πρόγραμμα επιτήρησης της ε, σπουγκόδους εγκεφαλοπάθειας και είναι σαφές επίσης ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση του ορίου ηλικία για τον έλεγχο των βοηδών θα είναι δυνατή μόνον εφόσον τα επόμενα χρόνια διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να μειώνονται οι περιπτώσεις διότι βεβαίως δεν είναι πολλές αλλά είναι 67 περιπτώσεις μέσα στο 2009 μια δεκαετία μετά από το αποκορύφωμα τότε της ε, κρίσεως της ε, σπογκόδους εγκεφαλοπάθειας. Επανέρχομαι τώρα στην απαγόρευση χορήγησης ζωικών πρωτεϊνών για τα οποία μίλησαν οι συνάδελφοι όπως και ο κύριος Νίκολσον, εγώ ποτέ δεν ήμουν υπέρ της απαγόρευσης χορήγησης ζωικών ε, πρωτεϊνών. Εγώ πάντοτε θεώρησα ότι είναι υπερβολικό, ότι είναι ακτιβισμός για να ικανοποιήσουμε κάποιες απόψεις της κοινή γνώμης. Έχει καλώ. Μπορεί αυτό να είχε και την θέση του κάποτε. Αλλά κάποια στιγμή οφείλουμε να δούμε ότι χρειάζεται να είμαστε ορθολογικοί. Και δεν υπάρχει κανείς λόγος για τον οποίο ζώα παμφάγα που πραγματικά τρώνε τα πάντα. Γι' αυτό και λέγονται παμφάγα. Γιατί τέτοια ζώα να μην μπορούν άραγε να φάνε ένα τμήμα άλλου ζώου το οποίο θα το έκαναν και αν ζούσαν ελεύθερα στην φύση. Διότι μιλάμε βεβαίως για κατάλοιπα σφαγής Μπορούμε να πούμε ίσως ότι ενοχλεί την αισθητική ή ότι δεν είναι ωραία πράγματα, αλλά τέλο πάντων αυτά είναι όντως ζωικές προτείνει, ζωικό λεύκομα. Είτε λοιπόν, ε, ε, ε, μάλλον έχουμε το δικαίωμα να τα σπαταλάμε τα πράγματα αυτά, δεν ξέρω. Ο Τζιμ Νίκολσον είπε ότι κατανοεί την πίεση που ασκεί η κοινή γνώμη. Ή την οικονομική πίεση μάλλον εγώ αμφισβητώ ότι είναι καν και ηθικό το να σπαταλάμε τα τμήματα αυτά των ζώων, να μην τα χρησιμοποιούμε δηλαδή. Και θεωρώ, όπως θεωρούσα και παλαιότερα, ότι οφείλουμε να το κάνουμε. Δέχομαι τα όσα περιέγραφε στην έκθεσή της η κυρία Πάουλσεν περί κανιβαλισμού προετών και σε άλλες εκθέσεις που έκανε μετά η κυρία Πάουλσεν και ο κύριος Συνεργάτη. Το δέχομαι, και το σέβομαι. Η κυρία Πάουλσεν ρώτησε πώς μπορεί να διαπιστώσει κανείς από ποιο ζώο προέρχεται το ε, συγκεκριμένο υλικό. Η Κομισιόν θα πει βέβαια σχετικά σε λίγο, αλλά υπάρχουν μέθοδοι που το καθιστούν αυτό δυνατό και που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μέθοδοι αυτοί και που κρύβονται πίσω από την μέθοδο PCR θα τα πούνε οι εκπρόσωποι της Κομισιόν σε λίγο. Πάντως αυτές οι δυνατότητες έρευνας υπάρχουν το δεύτερο εξάμεινο του 2011 και εγώ γράφω στην έκθεσή μου ότι η άρση της απαγόρευσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή αξιόπιστης μεθόδου για την ε, διαπίστωση του πόθεν προέρχονται οι συγκεκριμένες ζωικές πρωτεΐνες. Τώρα τι γίνεται με τα όρια ανοχής. Εγώ δεν είμαι ιστερική σε τρόπο που να πω ότι μυρικαστικά τα οποία τρώνε βεβαίως μόνο ε, χόρτα δεν θα φάνε και ένα σκουλικάκι το οποίο κυκλοφορεί πάνω στα χόρτα. Βέβαια θα το κάνω αυτό. Τώρα, η εγκεφαλοπάθεια στα ζώα δεν προέρχεται από αυτό. Ασφαλώς προέκυψε, δεν ξέρω από εκείνα από, εκείνους, από εκείνα, ε, ε, ε, εκείνους τους ιούς που προήλθαν από τους εγκεφάλους, εγκεφάλους ε, άρρωστων προβάτων. Δεν μιλούμε για τον ποντικό που ενδεχομένως θα πέσει κάποια στιγμή μέσα στο, ε, στην ε, προέλευση ζωοτροφή. Υπάρχουν βεβαίως ήδη κάποιες ρυθμίσεις για όρια Αντοχή για το ποντίκι που έπεσε μέσα ή το πουλί ή δεν ξέρω τι. Έχουμε μιλήσει για την ανικιοθελή ε, μόλυνση αλλά να υπάρχει τώρα οριακή τιμή και για το κρέας ζώων στις φυτικές πρωτεΐνες. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε, διότι αυτό θα ήταν ασφαλέστατα λάθος μήνυμα. Δεν μπορούμε, δεν επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό. Και Βεβαίω γνωρίζετε ότι γενικά είμαι ανοιχτή σε συμβιβασμού, αλλά αυτό δεν μπορώ να δεχθώ να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, τέλος πάντων ας μπει και λίγο ζωικό άλευρο, δηλαδή ζωική προέλευσης σε ε, τροφές για αγελάδε. Τώρα ο κ. Σνέρχαρτ είπε επίση ότι είναι κατά της φαγής της αγέλη. Γνωρίζουμε ότι εφόσον σε μια αγέλη υπάρξει μια περίπτωση σπογκώδους εγκεφαλοπάθεια, είτε θανατώνεται ολόκληρη αγέλη και απαγορεύεται η χρήση του κρέατό του, είτε η χώρα μέλο υποβάλλει αίτηση να επιτραπεί στα ζώα να ζήσουν μέχρι τέλους τη παραγωγικής του ζωή για την παραγωγή γάλακτος ή δεν ξέρω τι. γάλακτο η Ευρωπαϊκή πουμε τωρα όπω ότι υπάρχει, θα υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουμε κατά τα ιωθώτα και να πούμε, ε, τέλος πάντων, μία περίπτωση σπογγόδους εγκεφαλοπάθειας. Εντάξει, θα εξετάσουμε και τα υπόλοιπα ζώα post-mortem βεβαίως. Αυτό, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Το θεωρώ, για να είμαι ειλικρινής, πώς να πω, το θεωρώ ε, παράτολμο, προκλητικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ασφαλώς κάτι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα το δεχθεί αυτό η κοινή γνώμη. Ας υποθέσουμε μια αγέλη ε, σε, σε ένα λιβάδι στη Γερμανία. Ωραία. Και συνεχίζει τη ζωή της απρόσκοπτα και χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό για μένα είναι αδιανόητο. Και στην πράξη δεν παίζει και ρόλο. Εφόσον μια χώρα μέλος θεωρήσει ότι επιθυμεί να διατηρηθούν τα ζώα εν ζωή μέχρι τέλους της παραγωγικής του ζωής, αυτό έχει καλώς. Αλλά να μπουν τα ζώα στην παραγωγή του κρέατος, εν τέλει, αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι απολύτως αδικαιολόγητο. 67 περιπτώσεις το έτος 2009. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπει. Ας τα ξαναπούμε ίσως το 2013, 2014, 2015, όταν ίσως να έχουμε τρεις περιπτώσεις. Κρούσματα εννοώ δηλαδή. Τρία κρούσματα ή δύο έστω. Θα δούμε τότε γιατί εγώ θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ λάθος ως μήνυμα. Ο κύριος Σνέρχαρτ μίλησε πάλι για την διοξίνη. Εγώ δεν μιλώ για την διοξίνη που εκπέμπεται τυχαία στα ε, λιβάδια, αλλά για την διοξίνη στα ηχθιάλευρα, που είναι τεχνητό το όριο. Τα έχω πει παλαιότερα και στους επιτρόπους Φίσλερ και άλλους. Δεν έχουν ληφθεί εκεί τα, υπόψη τα κριτήρια της ε, προστασίας της ανθρώπινης υγείας, αλλά μόνο για να μπορέσουν να προστατευτούν κάποιες αλίες μικρών λευκών ψαριών από τη Βόρεια Θάλασσα. Πρέπει λοιπόν να επανεξεταστεί το θέμα της διοξίνης και ιδίως εάν το ηχθιάλευρο με υψηλότερο ποσοστό διοξίνης από ό,τι μέχρι τώρα μπορεί να χορηγηθεί ως λεύκομα, ιδίως στα πουλερικά και μήπως αντιθέτως θα πρέπει να μειωθεί το όριο ανοχή. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η επανεξέταση είναι απαραίτητη. Τώρα, επίσης, Σνέλχαρτ και Πάουσεν αναφέρθηκαν στην παράγραφο 22 για τι εγκαταστάσεις βιοαερίου. Μετά από 14 χρόνια που ασχολούμαι με την ε, σπουγόδη κεφαλοπάθεια και έχω προεδρεύσει και της ε, αρμόδιας τότε υποεπιτροπής, Έχω μιλήσει με πολλούς και ευρωβουλευτές και πρώην ευρωβουλευτές, οι οποίοι μάλιστα είναι και αγρότες και ένας μάλιστα που ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας τότε, μου τόνισαν και πάλι, και γι' αυτό το περιέλαβα αυτό, το 22, ότι πρέπει να έχουμε κάποια συνέπεια σε ό,τι αφορά την υγιεινή των υποπροϊόντων των ε, ζώων. Ε, γι' αυτό μου είχε πει ο κύριος Τσουμπάρινγκτορ τότε, εφόσον έχουμε αυστηρούς όρους για την χρήση των ζωικών αλεύρων και για την αποστήρωσή τους, το ίδιο πρέπει να έχουμε εφόσον το υλικό αυτό κατευθύνεται και σε εγκαταστάσεις βιοαερίου, που ενδεχομένως να έχει δυσμενείς επιπτώσεις μέσω των αερίων καύσεως σε ε, γειτονικά λιβάδια. 70 λοιπόν βαθμοί τουλάχιστον Κελσίου για την ε, ε, επεξεργασία των υλικών αυτών. Η κυρία Πάουλσεν μίλησε πάλι για την απαγόρευση του κανιβαλισμού. Εγώ την υποστηρίζω την απαγόρευση αυτή. Αυτή αναφέρθηκε στην παράγραφό μου υπαριθμών 20 που αναφέρεται πάλι και στις διοξίνες και εκεί έχω γράψει εγώ κάτι για τους ε, κανόνες ελέγχου. Οι έλεγχοι τροφίμων βεβαίως προβλέπονται από την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από εκεί πέρα η εφαρμογή είναι θέμα των χωρών μελών. Αυτό το επαναλαμβάνω εγώ στην συγκεκριμένη παράγραφο, ότι δηλαδή οι χώρε μέλη καλούνται να ελέγχουν αυστηρά τα επίπεδα διοξίνης και ενδεχομένως και να επιβάλλουν και αυστηρότερους κανόνες. Γιατί σε σχέση με τις ε, υποθέσεις διοξίνης έχουμε διαπιστώσει ότι οι χώρες μέλη σπανιότατα ελέγχουν τις διοξίνες. Ελέγχουν τα πάντα, αλλά όχι τις διοξίνες. Και γι' αυτό περιέλαβα την παράγραφο 20. Για τον Τζιμ Νίκολσον τώρα. Αναφέρθηκες σε μια ανησυχία σχετικά με την διατήρηση της απαγόρευσης χορήγησης. Παρ' όλα αυτά θεωρώ, Τζιμ, ότι τώρα θα πρέπει να την άρουμε την απαγόρευση αυτή. Θαυμάσια είναι τα συναισθήματα των διαφόρων, αλλά εδώ δεν πρέπει να υπερισχύσουν. Το να μην χρησιμοποιούνται πρωτεΐνες από υπόλοιπα σφαγίων, ε, σφαγίων το γη δηλαδή, είναι λάθος. Έχεις δίκιο ε, στο εξή ότι είναι θέμα συναισθηματικά φορτισμένο, το γνωρίζω. Και γνωρίζω ότι η συναισθηματική φόρτιση υπάρχει και εδώ στην Ευρωβουλή. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και νομίζω ότι η ειλικρίνεια είναι ο καλύτερο ε, καθοδηγητή μα. Τμήματα του χειρίου, ή, του χειρινού μάλλον ή του πουλερικού μπαίνουν και στο στην διατροφή του κατοικιδίου. Προτιμάμε να πεταχτούν και ταυτόχρονα να αγοράζουμε σόγια γενετικά μεταλλαγμένη ή μη στην παγκόσμια αγορά. Και πάλι και αυτό δεν είναι επαρκής πηγή ε, Πρωτενη για τα ζώα. Χρειαζόμαστε, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα πρωτενή και χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο. για το μηχανικά διαχωρισμένο κρέα εγώ θα προτιμούσα να απαγορευτεί. Αυτό ε, βεβαίω δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Είναι ζήτημα των χωρών μελών. Και για τη σόγια τώρα, πάλι, η σόγια βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο στην τροφική αλυσίδα. Και κυρίως για τα μη παμφάγα. Το γνωρίζω, αλλά δεν είναι και το μοναδικό και δεν έχουμε και αρκετά, αρκετές ε, ε, καλλιέργειες ε, ελαιοδών φυτών και εν τέλει τα χρησιμοποιούμε και για βιοκαύσιμα. Καλά, έστω, τα φυτεύουμε και τα βάζουμε μετά στα αυτοκίνητά μας. Κάπου πρέπει να βάλουμε και ένα όριο. Αυτό πρέπει να το πούμε επίσης στον κόσμο, Jim. Ε, εφόσον όμως κύριοι καταναλώνετε κρέας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ζώα αυτά, τα σφάγια αυτά όλοι θέλουμε να ζουν μια υγιή, υγιή ζωή, να βρίσκονται βεβαίως έξω και τα λοιπά, αλλά χρειάζονται να φάνε. Και όσο περισσότερο ζουν, τόσο περισσότερη τροφή χρειάζονται. Και βεβαίω αυτό θέλουμε. Τουλάχιστον σε ορισμένε ε, χώρες μέλη, ιδίως στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο, βέβαια και στη Γερμανία ιδιαίτερα. Ό,τι είδους σόγια και να χρησιμοποιήσουμε δεν μας αρκεί γενετικά τροποποιημένη μία. Έχει λοιπόν καλώς, σας ευχαριστώ. Είμαι βεβαία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να μας φωτίσει και εγώ την αναμένω με μεγάλη υπομονησία. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πούτλε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Ε, με ιδιαίτερη χαρά ερχόμαστε εδώ 25 χρόνια μετά το πρώτο κρούσμα που διαγνώστηκε το 1986 στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια ακόμα έκθεση της κυρίας Ροτ Μπέρεντ. Και πολύ δε περισσότερο χαιρόμαστε που η έκθεση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα επικριτική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενικά Είμαστε πάρα πολύ υπέρ των προτάσεων της Ευρω... Ε, κυρίας Ροτμπέρεντ και των συμπερασμάτων της. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις μπορώ να απαντήσω ε, συντομία μια επισκόπηση των διαφόρων θεμάτων για την εποπτεία και την παρακολούθηση. Βεβαίως ε, προτείναμε μέτρα για να μειώσουμε τον αριθμό των δοκιμών και να αυξηθεί η ηλικία, αλλά θέλουμε να Υπάρχει ένα σύστημα που να παρακολουθεί την επίπτωση ε, της ασθένειας, ε, κρούσματα και σε ζώα που ε, πεθαίνουν στην εκμετάλλευση είναι η ύποπτα. Για 67 περιπτώσεις μίλησε η κυρία Ροτ Μπέρεν το 2009, 35 περίπου το 2010. περίπου κάθε χρόνο μειώνεται στο μισό αριθμό των κρουσμάτων και ελπίζουμε να φτάσουμε στο μηδέν. Ε, κάποια στιγμή ή αρκετά περιορισμένο. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και αυθόρμητες περιπτώσεις εκφυλισμού του εγκεφάλου που μοιάζουν με σπογκώδη κεφαλοπάθεια και δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε ακριβώς και να τις ανιχνεύσουμε. Αλλά οι περιπτώσεις που μεταδίδονται με ζωικά άλευρα έχουν τερματιστεί τελείως και ακόμα θετικές ε, περιπτώσεις τα κρούσματα ή τα περιστατικά είναι ζώα που έχουν ε, μολυνθεί προδεκαετίας και πλέον. Και είναι γεγονό ότι αποτελεί όνειρο για όλους μας να έχουμε ε, δοκιμές ε, στο ζώο, ε, ante mortem, δηλαδή όχι η νεκροψία του εγκεφάλου με ένα τρόπο ανάλυση βιολογικών ιστών ή με μια εμολυψία. Συγγνώμη. Αλλά αυτό ε, είναι όνειρο γιατί οι ερευνητές δεν μας ε, δίνουν ελπιδοφόρα μηνύματα προς την κατεύθυνση αυτή. Για την απαγόρευση τώρα χορήγηση ορισμένων ζωοτροφών. Συμφωνούμε με τα συμπεράσματα της εισηγήτριας. Είδατε τον οδικό μας χάρτη ότι δεν τίθεται θέμα να προτείνουμε τα μη ρικαστικά να τρέφονται με ζωικά άλευρα. Ζούμε ε, ε, υπό το φάσμα του, της ε, ΣΕΒ ε, της δεκαετίας του 90 που είχαμε και, μέχρι και 30.000 κρούσματα το χρόνο. Δεν θέλουμε να ξαναφτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Επίσης επιβεβαιώνω αυτό που είπε η κυρία Ροτ Μπέρεντ, δηλαδή ότι τα ε, ερευνητικά εργαστήρια γύρω στα τέλη του 2011 θα είναι σε θέση να μας υποβάλουν ε, δοκιμές PCR ε, για να ανοιχνεύουμε στα άλευρα αν υπάρχουν ζωικές πρωτεΐνες και από ποιο είδος. Ακριβώς για να μην έχουμε διασταυρωμένη ε, διατροφή, δηλαδή να δίνουμε πουλερικά στους χείρους και χείριο ε, λεύκομα στα πουλερικά, χρειάζονται δοκιμές. Δεν μπορούμε έτσι στα τυφλά και θα το υποβάλουμε και ε, στην κρίση και στην απόφαση του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Βεβαίω οι εισαγωγές επίσης θα ελέγχονται έτσι ώστε να βεβαιωνόμαστε ότι αυτές οι μαγικές παράμετροι 133 βαθμοί, 20 λεπτά και 3 μπαρ ε, να ε, τηρούνται ως προδιαγραφές ε, επεξεργασίας των αλεύρων που εισάγονται από τρίτες χώρες. Για το υλικό ειδικού κινδύνου, επίσης δεν τίθεται θέμα να ευθυγραμμιστούμε στο Διεθνές Γραφείο Επιζωτιών. Ακολουθούμε την ΕΦΣΑ εμείς, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων. Αν και πιστεύουμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βγει το έντερο το λεπτό έντερο. Γνωρίζετε σήμερα ότι θεωρείται υλικό ειδικού κινδύνου όλο το έντερο των βοηδών και καταστρέφεται. Ενώ από ό,τι φαίνεται οι προσβεβλημένοι ιστοί ε, αφορούν μόνο ένα μέτρο του ε, εντέρου από τα 15 που είναι το σύνολο στο βοηδή. Πάντως δεν είναι σαφή ακόμα τα μηνύματα από την ερευνητική κοινότητα και την επιστημονική, οπότε εφόσον δεν είμαστε 100% σίγουροι, καλύτερα να καταστρέφετε το 100% του εντέρου. Ε, πάντως είναι σημαντική απώλεια ε, σε τόνους υλικού. Για την έρευνα τώρα, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να βρούμε ε, γενετική αντοχή για τις ε, έγες. Ερώτησε ο κύριος Σνέλχαρτ για τα βοηδή, είναι λιγότερο σαφές. Για τα πρόβατα υπάρχει, για τα εγωιδή μπορεί κάποια στιγμή ε, να βρεθεί αυτή η γενετική αντοχή. Έχουμε εμπειρία στην Κύπρο ακριβώς επ' αυτού, αυτό τον καιρό και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν πιθανότατα το 2012. Για τα βοηθή δυστυχώς είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι όλοι θα ελπιζαν να έχουμε γενετική αντίσταση με δυνατότητα διασταύρωσης των ζώων κτλ. για να έχουμε ανθεκτικά γονίδια. Για τους επίσημους ελέγχους τώρα. Συμφωνούμε και με την κυρία Πόλσεν για τους διατροφικούς ελέγχους που δεν γίνονται ίσως με τρόπο εναρμονισμένο ή αρκετά εναρμονισμένο στα κράτη-μέλη. Είναι γεγονός. Οι συνάδελφοι από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων ελέγχουν όλη την τροφική αλυσίδα, όχι μόνο τι ζωοτροφέ για τη σπογκώδη κεφαλοπάθεια των βοηδών, φύτο υγειονομική, ε, την υγιεινή των τροφίμων, ε, όλη την τροφική αλυσίδα από το φυτό μέχρι ε, το ζώο, πώς θα τραφεί, πώς θα καταλήξει σε τρόφιμο. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα. Οι περισσότερες κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πολύ μεγάλες δυσκολίες ορισμένες, όπως είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Και δυστυχώ, η ένταση των ελέγχων στο κλάδο αυτό και σε όλη την τροφική αλυσίδα ε, πλήττεται. Πάντω γίνονται εκθέσεις, γίνονται αναφορές, καμιά φορά και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κατάρτιση που ονομάζεται στα αγγλικά Better, Better Training for Safer Food, καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα, καταφέρνουμε κάπως να βελτιώνουμε την κατάσταση και την εκπαίδευση. γιατί σε ΣΕΒ όμως, από την αρχή, θυμάστε ο Επίτροπος Μπέρν ε, το 2000, είχε ε, δώσει προτεραιότητα στο κτηνιατρικό γραφείο να ασκήσουν πίεση συγκεκριμένη για ελέγχου στα κρατη Και χάρη σε αυτό, για τη σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια των βοηθών, γενικά είχαμε ε, ε, αυστηρότερους ελέγχου για τα παλιά και πολύ ε, σφιχτούς. Για τις διοξίνες τώρα στα ηχθιάλευρα. Θα ήθελα να επιμείνω στο εξής. οι οριακέ τιμέ είναι πάρα πολύ αυστηρέ στα αλευρά για διοξίνε και μάλιστα οι του κόσμου. Τι αναθεωρήσαμε μετά από διάφορες επιστημονικές μελέτες ή εκθέσεις. Γνωρίζετε ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη Βαλτική ε, συγκεκριμένα. Πάντως, ε, είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα της ε, διοξίνης. Έχουμε επίγνωση ε, η κρίση στη Γερμανία πρόσφατα στα τέλη του 2010 και αρχές του 2011 μας ξανάφερε όλα αυτά τα θέματα στο προσκήνιο ακόμα και αν η προέλευση δεν έχει ξεκαθαριστεί από τη γερμανική δικαιοσύνη εξ όσο γνωρίζω ακόμα ε, πάντως είναι πάρα πολύ αυστηρές οι προδιαγραφές οι αυστηρότερες το δυστύχημα είναι ότι Υπάρχουν συστήματα ε, ορισμένων πρωτεϊνών στα ηχθιάλευρα συγκεκριμένα και στα ηχθή Μάλλον, στα ηχθή ναι, αλλά στα ηχθιάλευρα δεν μπορεί να απορρίπανθει, να αφαιρεθεί η διοξίνη από το αλεύρι. Από το ηχθή μπορεί. Ε, και εκεί έχουμε πρόβλημα. Αλλά γνωρίζουμε ότι τα ηχθιάλευρα ε, ως πηγή πρωτεΐνης είναι σημαντική. Ακόμα και αν σε επίπεδο έτσι, παγκόσμιο μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι ε, από πλευρά αηφόρου ανάπτυξης και αλλιευμάτων είναι πρόβλημα να ψαρεύουμε ψάρια για να ταΐζουμε ζώα. και στον οδικό χάρτη ε, το έχουμε προβλέψει, είναι ε, πολύτιμη ε, πηγή πρωτεϊνών, αυτό το είδος των αλεύρων, όχι για τα μυρικαστικά αλλά για άλλα είδη και καλό θα ήταν να τα χρησιμοποιούμε για να αποφύγουμε τις εισαγωγές γενετικά τροποποιημένης σόγιας από χώρες της Αμερικής, Βορείου και Νοτίου. Για τις αγέλες ή τις ομάδες ζώων που θανατώνονται, προτείναμε ένα σύστημα Όταν σε μια εκτροφή έχει ε, εντοπιστεί κρούσμα σε εγκεφαλοπάθης, να συνεχίζει το υπόλοιπα ζωά να υφίστανται εκμετάλλευση καθ' όλη τη διάκριση της ζωής του για τα προϊόντα τους και να μην θανατώνονται. Ας πούμε οι γαλακτοπαραγωγές αγελάδες δεν συνεχίζουν να παράγουν γάλα ε, διότι το, το, πρίον, το πρίον η πρωτεΐνη αυτή δεν μεταδίδεται με το γάλα και όταν τελειώσει ο γαλακτοπαραγωγικός τους βίος να διατίθενται σε ανθρώπινη κατανάλωση μετά από κατάλληλους ελέγχους. Αν πραγματικά υπήρχε πολιτική βούληση να μην ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να μην ολοκληρώνεται ο παραγωγικός βίος των ζώων με αυτόν τον τρόπο, αλλά να θανατώνονται και να ε, καίγονται, δεν θα υπήρχε πρόβλημα στο τέλος της ζωής τους όμως. Και αυτό αφορά λίγα ζώα γιατί όπως σας είπα μειώνονται συνεχώς τα κρούσματα και οι αγέλες αυτές. Για το μηχανικό διαχωρισμό του κρέατος. Ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα πολύ προσφυλές της κυρίας Ροντ Μπέρεντ. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τι είναι αυτό. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε αρχίσει μάλλον μια προσπάθεια μείωσης των ε, διατροφικών αποβλήτων. Ξέρετε ότι πετάμε πολλά τρόφιμα και τα καταστρέφουμε. Ενώ είναι ακόμα κατάλληλα για κατανάλωση. Αυτό είναι ένα θέμα και ένα πρόβλημα και ε, ως προς την ένδυα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εφορία και την ανακύκλωση. Είναι γεγονός ότι όταν ψάχνουμε και την τελευταία σάρκα που πρέπει να τη βγάλουμε από τα οστά, συνθλίβοντάς τα, με τεράστια πίεση για να ξεκολλήσει από το κόκαλο. Ε, αυτό δεν είναι πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, όλοι το αναγνωρίζουμε. Από την άλλη όμως είναι πρωτεΐνη που από πλευράς υγειονομικής ε, είναι κατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση. Όταν γίνεται με καλούς τρόπους και στα πουλερικά έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες για να αποφύγουμε τη μόλυνση με σαλμονέλα, ε, στους χείρους λιγότερο, αλλά και πάλι με πολύ συγκεκριμένες ε, προϋποθέσεις, τα βοηδή απαγορεύεται αυτό. Αλλά Αλλά παρόλα αυτά παραμένει πηγή πρωτεϊνών αυτό το υλικό. Και θα επιθυμούσαμε να αποφύγουμε απώλεια αυτών των πρωτεϊνών. Γενικά σε ένα ε, σφάγιο, ανεξάρτητα από το ζώο, 45% του σφαγίου ε, πηγαίνει σε ανθρώπινη κατανάλωση και 55% είναι είτε παραπροϊόντα που πηγαίνουν στην κατανάλωση των ζώων ή υποπροϊόντα ε, για κομποστοποίηση, παραγωγή λιπασμάτων ή ε, ε, καίγονται πλήρως υπολείμματα σφαγίων. Είναι υψηλό αυτό το ποσοστό, πάνω από το μισό σφάγιο έτσι, ενό ζώου, είναι 55%. Και αν μπορούμε μερικά ποσοστά έτσι να τα <laughs> ξύσουμε, και να δώσουμε στον καταναλωτή ένα κρέας όχι υψηλής ποιότητος μεν, αλλά ασφαλές, πρωτεΐνες, ζωικές, που γίνονται ελλαντικά. Γιατί όχι, να μην το σκεφτούμε και αυτό. Αν υπάρχει όμως η πολιτική βούληση απαγόρευσης ε, αυτό, του, του μηχανικού διαχωρισμού, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να υποκληθούμε σε αυτή. Έχει σημασία πάντως γιατί είναι και ένα τμήμα των εξαγωγών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αγοράζουν τρίτες χώρες που αγοράζουν ακριβώς αυτές τις πρωτεΐνες χαμηλότερη τιμή, αλλά στα πουλερικά όταν πρόκειται για τόνους είναι και σημαντική η οικονομία που γίνεται. Αυτά κυρία Πρόεδρε, ε, σχόλια από πλευράς μας. Και τέλος θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ροτ Μπέρεντ για την έκθεσή της και πάλι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Όλοι σας συγχαίρουν. Ε, μήπως η συγγήτρια θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Για να κλείσει σήμερα η συζήτηση, το μόνο που έχω να πω είναι ότι ευχαριστώ για τόσο χρόνο που είχαμε. Δεν είναι καθόλου προφανές στην Επιτροπή μας. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους σκιώδεις ηγητές, ειλικρινά, για την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω την άλλη εβδομάδα να μπορέσουμε να συγκαλέσουμε μία συγκέντρωση με τους σκιώδεις ηγητές. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Πουτλέ σε όλα, σε ό,τι αφορά τη θανάτωση ε, όλης της Αγέλης, ούτε με τον κύριο Σνέρχαρτ. να το κοιτάξουμε αυτό, πώς θα συνεννοηθούμε. Ε, Σω θα πρέπει να επανέλθουμε του χρόνου ή σε δύο χρόνια. Αν συνεχίσουν να μειώνονται τα κρούσματα, καλώς. Και ήδη σήμερα, κύριε Ποντελέ, οι γαλακτοπαραγωγέ αγελάδε δεν είναι υποχρεωτικό να θανατώνονται. Μπορούν να συνεχίζουν να παράγουν γάλα. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε την νομοθεσία. Μπορούμε να πούνε στα κράτη-μέλη να το ζητήσουν, να υποβάλουν ένα αίτημα. Εάν δεν το θέλουν, εάν δεν το επιθυμούν, δική του υπόθεση είναι. Συμφωνώ μαζί σα αυτό. Γενικά δεν συμφωνώ ε, με αυτό το κρέας, το μηχανικά διαχωριζόμενο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ε, όταν ε, είχε φουντώσει σπογκώδη κεφαλοπάθεια, υπήρχε κίνδυνος, ενδεχομένως κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, δεν το ξέραμε. Και είπαμε ότι να έχουμε μόνο κρέας από εμεί Και για μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι στις αγελάδες, μπορούσαμε και πουλούσαμε κρέας με το κόκαλο. Ε, η σπονδυλική στήλη δεν ήταν στο σύνολό τη υλικό υψηλού κινδύνου, ε, ανάλογα με την ηλικία ε, του ζώου. Σε ορισμένε χώρε είχαν απαγορευτεί οι μπριζόλε με το κόκαλο, T-bone, στην Ιταλία, πώ τη λένε, Φιωρεντίνα, εκεί πέρα την μπριζόλα τη μεγάλη. Και σε αυτό το μηχανικά διαχωριζόμενο κρέας πάντα ε, υπάρχει δυνατότητα τραυματισμού του οστού και όντως τραυματίζεται το οστό και βγαίνει και μυελό στο οστού. Ο κύριος Σνέλχαρτ λέει όχι. Μα είναι ευρεία πρακτική, κύριε Πούντελε, πραγματικά εξηγήστε στον κύριο Σνέλχαρτ ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Ότι ε, έχετε και φράσματα οστών πολύ συχνά. Μα είναι προφανές αυτονόητο, είναι καθημερινή πρακτική, οφείλουμε να το δεχτούμε, να το ξέρουμε. Κύριε Πούντελε, Εκτιμώ πολύ αυτά που λέτε για την αγορά και την Ευρώπη. Αν χρειαζόμαστε πραγματικά αυτό το μικρό ποσοστό και παίζει τέτοιο ρόλο για τις εξαγωγές, δεν μπορώ να τα δεχτώ αυτά και, να συμφωνήσω. Με τη σήμανση όμως να λέει, ε, όχι πολτοποιημένο, δεν ξέρω πώς το γράφει εκεί πέρα ε, στα λαντικά, αλλά να γράφει ε, ότι έχει παραχθεί από κρέα που έχουμε κερδίσει με μηχανικά μέσα ή κάτι άλλο, καταλαβαίνει ο κόσμος. Εκεί να δείτε πώς θα το αγοράζουν. Και να βάλουμε σήμαση για όλα αυτά που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, στην προστινή ε, πλευρά του, του τροφίμου που μας ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τότε θα λυθεί από μόνο του το πρόβλημα, διεκπαιρώνεται έτσι. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι θα πρέπει να στέλνουμε τα σκουπίδια μας και ζητώ συγγνώμη που το λέω έτσι ε, και να τα στέλνουμε για ανθρώπινη κατανάλωση. Να τα κάνουμε ζωικά άλευρα και αυτά τα ζωικά άλευρα φυσικά δεν είναι τα οστά, είναι τα υπολείμματα κρέατος και τα υπόλοιπα να τα πετάμε. Εγώ δεν μπορώ να απαγορεύσω ε, το μηχανικό διαγορισμό, αλλά θα ζητήσω πιο αυστηρούς κανόνες και σήμανση για να δω και τι επιχειρήματα θα ακούσω ότι δεν γίνονται αυτά. Ευχαριστούμε κυρία εισηγήτρια. Η προθεσμία είναι 19 ε, Απριλίου στις 12 η ώρα. Θα ξαναβρεθούμε στις 24 Μαΐου και ε, στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Σας εύχομαι καλό βράδυ.